Uh, good morning, everybody. I think um, we should Ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας πάρω το αριστερό μικρόφωνο για να φέρομαι πιο καλά. Όποιος ε, άνοιξε λοιπόν το διαδίκτυο και τον υπολογιστή του 9 το πρωί με βλέπετε, βλέπετε και την κυρία Κρούς που είναι δίπλα μου την καλωσορίσω. Έχουμε μια νέα επιστολή της ένα ε, νέο δελτίο μάλλον της Επιτροπής μας, το διανύμαμε. Θα δώσουμε και στην Επίτροπο το σχετικό αντίγραφο, αντίτυπο, που άλλωστε μπορείτε να παρακολουθήσετε και από το διαδίκτυο. Καλωσορίζω λοιπόν με χαρά την κυρία Νέλη Κρούς, μας ε, συνοδεύει τακτικά στο έργο μας, παρακολουθεί τις συνεδριάσεις μας, ε, προσωπικό συνεργάζομαι και εγώ τακτικά μαζί της, ιδιαίτερα σε θέματα ε, ψηφιακής αγοράς. Θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Αρίας που ιδιαίτερα ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά και την ε, κυρία Γκάλερ, την κυρία Φαχέν, Γκαλό, την κυρία Φαχέν, που ασχολείται με το ψηφιακό νέφος και θα έχετε, κυρία Κρούς, όπως φαντάζεστε, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από πολλούς συναδέλφους. Ονομάζεται διαρθρωμένος διάλογος τεχνικά η συνεδρίασή μας εν ώψη των μελλοντικών εξελίξεων. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε γενικά τα θέματα του μέλλοντος για τις εξελίξεις στην αγορά. Και πιστεύω ότι και εσείς θέλετε να ανοίξετε το πεδίο. Επομένω, μπορείτε να αισθανθείτε ελεύθεροι και να μην περιοριστείτε μόνο στα θέματα της ασφάλειας των πληροφοριών, που είναι το κύριο θέμα σας σήμερα, από ό,τι ξέρω. Γιατί έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στο πρόγραμμά σας για το ψηφιακό θεματολόγιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μάλκομ. Θα κάνω κάτι το ασυνήθιστο σήμερα. Δεν θα ξαφνιάσω τον πρόεδρο γιατί με ξέρει αρκετά καλά. Αλλά αντί να σας εκφωνήσω έναν λόγο που βεβαίως έχω ετοιμάσει με τον ε, κατάλογο των ψηφιακών θεμάτων, την πρόοδο, τα προβλήματα και το οποίο αποστέλω σε μια επιστολή στον Μάλκολμ σήμερα ώστε να σας το διαβιβάσει ο πρόεδρος σας, να σας την διαβιβάσει ο πρόεδρος σας θα ήθελα να φερθώ στο τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ήμουν στο αεροπλάνο πηγαίνοντα στην Αίγυπτο, όχι για διακοπέ πρέπει να επισημάνω, αλλά για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, συνεδρίαση, συνάντηση με αγωνιστέ των ανθρωπινών δικαιωμάτων και bloggers και εκπροσώπους των μέσων κοινωνική δικτύωση. Γιατί κυρίε και κύριοι, αν εμεί παραπονιόμαστε, για πηγαίνετε μια φορά εκεί, έστω και για μια μέρα. Η γραμμή του είναι δεν τα παρατάμε ποτέ, δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Και πρέπει να σας πω ότι με είχε εμπνεύσει αυτό η, η συνάντηση. Διάβαζα λοιπόν τον ε, λόγο μου, την ομιλία και συνειδητοποίησα κάτι. Και σκέφτηκα ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται πολιτική συζήτηση, γιατί εδώ το Κοινοβούλιο, το Σώμα είναι ένα χώρος πολιτικής συνάντηση και αντιπαράθεση. Και εγώ αυτή τη δουλειά θεωρώ ότι εκπροσωπώ από τη δική μου την πλευρά. Έτσι λοιπόν, Εάν θέλουμε μια ε, ουσιαστική αγορά των τηλεπικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση στα πολιτικά κυρίως θέματα. Και αυτό το απευθύνω σαν παρατήρηση προς ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα του τα μέλη. Ξέρω ότι εσείς βεβαίως είσαστε οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου με την σύνθεση της Επιτροπής σας, αλλά πέραν ημών απευθύνω το μήνυμα σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε το θεματολόγιο το ψηφιακό και την ε, κυβερνοασφάλεια που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά εγώ αυτό που θα σας πω σήμερα είναι όχι μόνο αυτά, ας κάνουμε κι άλλα, ας κάνουμε περισσότερα. Είναι τα διακυβεύματα που αντιμετωπίζουμε εσείς και εγώ κοινά. Γι' αυτό πείτε μου λοιπόν, μπορούμε μαζί να κάνουμε κάτι το ξεχωριστό από σήμερα μέχρι τις ευρωεκλογέ που έρχονται. Αυτό είναι το θέμα που θέλω να διερευνήσουμε σήμερα. Θέλω εσείς και εγώ μαζί να δείξουμε στον πολίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει πράγματα στη ζωή τους. Συζητούμε, κάνουμε κουβέντα για αποτελέσματα και εκεί ακριβώς θέλω να επιμείνουμε στα αποτελέσματα, στην υλοποίηση των υπεσχημένων. Και θέλω καν... οι κανόνες για την ψηφιακή κοινωνία, την ψηφιακή τεχνολογία να αντιστοιχούν στα μελήματα και τις ανησυχίες των πολιτών. Ε, όπου ακούω να μιλάνε πολίτες στην Ευρώπη, αυτό που λένε πάντα είναι «Ναι, καλά μας τα λέτε, το καταλάβαμε αυτό με την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, το καταλάβαμε αυτό με την εσωτερική αγορά, αλλά σας παρακαλούμε, έχουμε κι εμείς θεμητές προσδοκίες και θέλουμε να μας δώσετε αποτελέσματα». Αυτά λέει ο πολίτη. Και θέλω ε, εσείς να μπορέσετε, και αυτό το λέω όχι ε, λόγω της ηλικία μου, επειδή είμαι πιο ηλικιωμένη από εσά, αλλά επειδή έχω και την εμπειρία μου στο παλιό καιρό από τα καθήκοντα που είχα σε εθνικό επίπεδο, θέλω να μπορείτε να πάτε στις εκλογικές σας περιφέρειες, ευρωπαϊκές εκλογικές σα περιφέρειες και να μπορείτε να πείτε στον πολίτη εμείς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της διαμετακόμισης στην κινητή τηλεφωνία. Και μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ουδετερότητα του διαδικτύου. Και μπορούμε εμείς, και το έχουμε πράξει, έχουμε αναλάβει πραγματική δράση κατά του κυβερνοεγκλήματος και κατά των λοιπόν ε, απειλών. Τώρα, 8,5 χρόνια που συνεργαζόμαστε, πολλοί από σας, ε, ίσω και σε άλλου τομεί, αλλά πάντως περισσότεροι από εσά με γνωρίζετε, καλά και δεν νομίζω ότι είμαι περίπλοκη, μπορεί να με καταλάβει κανείς εύκολα, είμαι Ολλανδή, τα λέω στα ράτα, δεν ξέρω από διπλωματίες και θα φαντάζεστε βέβαια ότι κάποιος και στην ηλικία μου δεν αλλάζει και εύκολα, ούτε και θέλω άλλωστε να αλλάξω. Και ξέρω ότι πάντοτε ε, έχουμε συνομιλήσει χωρίς όμως να συμμεριζόμαστε τις ίδιες γνώμες, την ίδια γνώμη πάντα σε διάφορους τομείς. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι με εντυπωσίασε βαθύτατα και αυτό σας το λέω εκ βάθους καρδίας η θέση του Κοινοβουλίου η δική σας η επιτροπή, της Επιτροπής σας Μάλκολμ εκεί όπου θέξατε το ζήτημα των δεσμεύσεων για τα ευρύτερα ψηφιακά θέματα στις οποίες δεν έχουμε φέρει αποτέλεσμα. Και εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι δώσατε το έναυσμα κατά τρόπον ορατό, αγωνίζεστε, συνεχίσατε να αγωνίζεστε για αλλαγές εκεί που πολλοί από τους ηγέτες ή δεν ήθελαν να ακούσουν ή δεν ήθελαν να καταλάβουν ή δεν ήθελαν να ασχοληθούν και αυτό πρέπει να πω ότι με επηρέασε θετικά. Μου δώσατε δηλαδή περισσότερο κουράγιο για αγώνα και γι' αυτό θέλω να ε, γίνω κοινωνός της γνώσης σας και κοινωνός του πάθου σας για να προχωρήσουμε στην νομοθεσία που χρειάζεται προκειμένου να υλοποιηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά. Όπου βρεθώ και όπου μιλήσω, εξηγώ ότι το πετράδι του θέματος της Ευρώπης είναι η ενιαία αγορά και αυτήν πρέπει να προωθήσουμε. Υπάρχει μια εσωτερική αγορά με τις ελλείψεις της, αλλά πάντως υπάρχει. Και η πεποίθησή μου, Μάλκολμ, είναι ότι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα με ένα πλήρες πακέτο, ένα ολόκληρο πακέτο μέχρι το Πάσχα του 2014 για τα ψηφιακά. Για φανταστείτε λοιπόν να το καταφέρουμε αυτό. Αλλά απαιτείται βέβαια στενή συνεργασία και απαιτείται οπωσδήποτε πολύ μεγάλη βούληση να καταλήξουμε στο στόχο αυτό ασφαλώς θα είναι κάτι πολύ καλό για την Ευρώπη, αν αμφιβολά. Οπωσδήποτε θα είναι πολύ καλό για την ε, οικονομία, θα δώσει νέα όθηση και θα καταρρύψει φραγμούς. Αλλά επίσης στο ψηφιακό θεματολόγιο εγώ βλέπω τον άνθρωπο περισσότερο και όχι τον, τους αριθμούς. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο μα κατηγορούν πολύ συχνά, ότι εμεί στι Βρυξέλλε δεν σκεφτόμαστε τον άνθρωπο. Εγώ σα διαβεβαιώ ότι σε αυτήν την περίπτωση τον άνθρωπο έχω υπόψη μου στο σχεδιασμό του θεματολογίου για την ε, κοινωνία τη πληροφορία και όχι του αριθμού. Για να κοιτάξουμε λοιπόν τη νέα γενιά. Εγώ από τους νεαρούς του, συμβουλίου ε, που με περιστοιχίζουν ε, έχω διδαχθεί πολλά. Είναι νέοι αλλάζουν ίσως πολύ συχνά, αλλά από την άλλη έχουν και το πλεονέκτημα ότι δεν ε, ε, κολλάνε σε μια ιστορία ή σε μια ε, δήλωση, σε μια βεβαίωση που θα τους χορηγηθεί χωρίς να την αφισβητήσουν. Και οι νέοι αυτό που ζητούν πάνω απ' όλα είναι η σύνδεση, η διασύνδεση, το να παραμένουν συνδεδεμένοι και εδώ ακριβώς αυτοί που μένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο περισσότερο είναι και η γενιά η οποία ψηφίζει λιγότερο. Είναι οι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν λιγότερο. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη λοιπόν. Και αφού μιλούμε για εμπλοκή όλων των πολιτών, πρέπει σε αυτούς να στραφούμε. Αυτοί λοιπόν θέλουν την ε, νέα, ε, τη νέα αυτή γενιά με ε, τη δυνατότητα να ξεφύγει από την ανεργία χάρη στην κοινωνία την ψηφιακή. Το συζητήσαμε πρόσφατα, Μάλκολμ, ότι η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή είναι τα φρικτά νούμερα της ανεργίας των νέων σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά πέραν των ε, λίγων αυτών κρατών μελών που έχουν πολύ κακά στοιχεία για την ανεργία, πρέπει να πούμε ότι κανένα δεν είναι στο απειρόβλητο της ανεργίας των νέων. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά το πρόβλημα, ιδάλλως θα μιλάμε για μια χαμένη γενιά με πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να ξεφύγουν από την ε, παγίδα της ανεργίας με μια καλή ψηφιακή κοινωνία και οικονομία. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και η πιο ηλικιωμένη γενιά σου, την οποία θα πρέπει να εξηγήσουμε κάπως περισσότερο, γιατί εσείς είσαστε ενήμεροι φυσικά, το ξέρω, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην ηλικία, χρειάζονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες για να παραμένουν σε καλή υγεία, σε καλή ε, ε, δράση στη ζωή και χωρί να χάσουν την αξιοπρέπειά του. Βλέπετε το βραχιόλι που φοράω, δεν θα σα πω ποια εταιρεία είναι, αλλά είναι ένα βραχιόλι το οποίο επαληθεύει ότι, όλη, ότι κάθε μέρα έχω ασκηθεί αρκετά. Έχω κάνει αρκετή σωματική άσκηση. Βλέπετε ότι δεν έχω ακόμα συμπληρώσει το, το μερίδιό μου σωματικής άσκησης σήμερα. Αυτό λοιπόν για μένα επαληθεύει, ελέγχει το τι κάνω για το σώμα μου, τι κάνω για τη φυσική μου κατάσταση. Και αν όταν φτάσει το, μέρος, το τέλος της ημέρας και δεν έχω συμπληρώσει ε, την ποσόστοση θα κάνω ακόμη ένα γύρο τετραγώνου τρέχοντα. Μην μου πείτε, με ρωτήσετε βέβαια αν αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και οικονοποίηση, αλλά πάση το κάνω. Πολλά λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά και πολλά διακυβεύονται και για την πιο ηλικιωμένη γενιά, στην οποία μπορούμε να προσφέρουμε την αξιοπρέπεια του να ζουν πιο μεγάλο διάστημα, πιο πολλά χρόνια, αλλά με καλή υγεία, να μένουν δραστήριοι και να έχουν και την φροντίδα που χρειάζονται, χάρη και σε αυτέ τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Και έτσι, εάν καταφέρουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε και την ψηφιακή διασύνδεση προ όφελο ακόμη και των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Το ψηφιακό μέρισμα, λοιπόν, μπορεί να φέρει και την κοινωνική συμμετοχή. Η συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο φέρνει και την κοινωνική ενσωμάτωση. Εγώ δεν λέω ότι έχω να σας δώσω την πανάκια που θα σας λύσει όλα τα προβλήματα και τις απορίες. Δεν μου το επιτρέπει και η ηλικία μου. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει να κάνουμε μια πρόταση η οποία θα είναι ισορροπημένη, η οποία θα είναι λογική και η οποία θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε και σύντομα σε αποφάσεις. Και έτσι, εδώ θα πρέπει και να αυτοπεριοριστούμε και εγώ και εσείς και εμείς ε, γιατί καλό είναι να γίνει συζήτηση, αλλά όταν τελειώσει ο χρόνος για τη συζήτηση, καλό είναι να έχουμε αποτελέσματα και εφαρμογή. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι το επόμενο δωδεκάμινο, ενώπιση των ευρωεκλογών, θα το αφιερώσω στην οικοδόμηση ε, γεφύρας μαζί με εσά, μαζί με τον πολίτη και την ψηφιακή κοινωνία. Είτε πρόκειται για την αγορά ενός εισιτηρίου για το τρένο, είτε πρόκειται για συναλλαγές, είτε πρόκειται για ε, ψυχαγωγία χρειάζεται να έχει ο κόσμος, ο πολίτης, αυτή την πρόσβαση και από το κινητό του τηλέφωνο και βέβαια όλοι θέλουν τον περιορισμό του κόστους της περιαγωγής. Είναι ένα από τα λίγα στα οποία ακόμη και πιο γκρινιάριδες θα συμφωνήσουν ότι η Ευρώπη τα έχει καταφέρει αρκετά καλά. Και αν θυμάστε τι ήταν ένα από τα ποιο ήταν ένα από τα πρώτα αποτελέσματα όπου ε, πήρε εύσημα η πρώτη Επιτροπή Βαρόσο, αυτό ήταν το θέμα της περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία. Φυσικά έκανε πολλά άλλα καλά πράγματα, αλλά αυτό ήταν το πρώτο. Και αυτό θα το είχαμε καταφέρει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μεγάλο βήμα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί για μας μια επιπλέον πρόκληση. Και αν μου δώσετε την ευκαιρία θα σας εξηγήσω. Γιατί έχω σαν χαρτοφυλάκιο θέματα που είναι ακριβώς στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης πολιτικής για την Ευρώπη, για την ιστορική αγορά. Και θα πω ότι όταν συζητούμε δεν μιλάμε εσείς και εγώ ή εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μιλάμε ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε να κρατήσουμε το πιδάλιο γερά μαζί και πρέπει να προωθήσουμε και άλλα θέματα των τηλεπικοινωνιών, του ψηφιακού θεματολογίου, ε, και να τα προωθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με προτεραιότητες. Αυτή είναι η ευθύνη η δική σας, η δική μου. Μια ευθύνη η οποία δεν είναι πάντοτε ε, εύκολη. Δεν σημαίνει πάντα εύκολες επιλογές, γιατί κάποια θέματα θα πρέπει να βγουν από το συνολικό πακέτο. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος να αλλάξει αυτό είναι μια ισχυρή ενιαία αγορά, μια γυρή ενιαία αγορά. Και αυτό μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι η Ευρώπη τα καταφέρνει στα ψηφιακά και να πούμε στο ψηφοφόρο ότι η Ευρώπη ακούει. Οι τηλεπικοινωνίες εγγίζουν κάθε σημείο της ζωής. Ο χρήστης ε, αναπτύσσει τεράστιες προσδοκίες από τις τηλεπικοινωνίες για κάθε κομμάτι της ζωής του. Και χθες είχα μια συνάντηση με υπουργούς ε, θεμάτων επιστημών τεχνολογίας αλλά και εκπροσώπους ε, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας με τα πιο μεγάλα κεφάλια που μιλούσαν για την ηλεκτρονική σύγχρονη τεχνολογία και δεν θέλω να επισημάνω πόσο εντυπωσιακά ήταν τα όσα μέσα σε ένα χρόνο επετεύχθησαν και ήταν όλοι αυτοί ε, πριν από ένα χρόνο, ε, ο ένας αντιμέτωπος με τον άλλον, αντίθετοι και πολέμοι ο ένας με τον άλλον, και μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε να τους φέρουμε κοντά, να τους εξασφαλίσουμε ένα πνεύμα συνεργασίας, να μην βλέπουν ένα τον άλλον σαν αντίπαλο και ανταγωνιστή. Και έτσι εχθές μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια μεγάλη συμφωνία για τα ηλεκτρονικά και το 10% στην παγκόσμια συμμετοχή μας στο, στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια αγορά που θέλουμε να αυξήσουμε σε 20% πάρα πολύ γρήγορα μέχρι το 2020 με την αντίστοιχη ανάπτυξη βέβαια και των θέσεων εργασίας που συνοδεύει αυτή η παρουσία οι τηλεπικοινωνίε δίνουν τόσο πολλές δυνατότητες, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Οτιδήποτε και να χρησιμοποιήσετε πλέον έχει διασύνδεση τηλεπικοινωνία. Και πρέπει να λειτουργήσουν βεβαίω οι αγορέ, πρέπει να λειτουργήσουν τα δίκτυα, πρέπει να γίνουν... Πρέπει να λειτουργήσουν τα μηχανήματα ασφαλώς και πρέπει να γίνουν και οι σχετικές επενδύσεις για να μην έρθει η ώρα που θα έρθει είτε η νέα γενναία ούτε οι πιο ηλικιωμένοι να μας πούνε για ένα λεπτό. Εμείς αγοράσαμε όλα αυτά μηχανήματα που τάχα θα μας ευκόλυναν τη ζωή και τελικά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα και ουσία. Αυτό θα το πληρώσουμε αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα περιτά, αμέτρητα, περιτά και άχρηστα προσκόμματα στην διασύνδεση. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το σκεφτόμουν ερχόμενοι στη συνεδρίαση. Γιατί είσαστε υποψήφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι στι εθνικέ εκλογέ. Αν μου επιτρέψετε, θα δώσω την απάντηση στη θέση σας ή θα προσπαθήσω να καταλάβω τις δικές σας προθέσεις σε ένα βαθμό γιατί δεν σας άρεσαν τα τεχνητά όρια, σύνορα. Και είπατε όχι, θέλουμε να τα ξεπεράσουμε. Σε ένα βαθμό γιατί θεωρήσατε ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα εάν η ελευθερία και ο ανταγωνισμό ε, αναπτύσσονται σε ευρύτερο πεδίο, αν έχουμε περισσότερε ελευθερίε και ανθρώπινα δικαιώματα πιο ουσιαστικά. Και εσύ, Μάλκομ, είσαι ένα από τα απτά παραδείγματα. Άφησε τι εθνικέ ε, ευθύνε και αρμοδιότητε στην ε, χώρα σου για να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πότε πότε καλείσαι και να δώσει εξηγήσει εκεί, φαντάζομαι, στην εκλογική σου περιφέρεια. Αλλά ε, στις τηλεπικοινωνίες, σε όλους τους τομεί πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για σύνορα, για όρια. Είναι ούτω ή άλλω τεχνητά αυτά και εξορισμού οι τηλεπικοινωνίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ονομάζουμε το δίκτυο παγκόσμιο δίκτυο World Wide Web ε, και δεν υπάρχει άλλο τομέα, αυτής της ατελούσας του Ευρωπαϊκή ενιαίας αγορά, που να είναι τόσο περιτά, τόσο άχρηστα αλλά και τόσο υψηλά τα εμπόδια και τα προσκόμματα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι έχει έρθει η ώρα πλέον να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι αργά, υπερβολικά αργά. Πρέπει όμως να έρθει η αλλαγή τώρα από κάθε πλευρά. Αλλά για να είμαστε ειλικρινεί. από εμά θα ξεκινήσει. Από αυτήν εδώ την αίθουσα, όπω είπε, θα ξεκινήσει το κίνημα, γιατί είναι ένα κίνημα. Και ελπίζω σε λίγο να έρθει η μέρα που θα αποκαλέσουμε τη σημερινή ημέρα, την 30η Μαΐου, η μέρα της μεγάλης στροφής στην ψηφιακή κοινωνία για την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι εμείς θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ε, διατύπωση ενός μεγάλου ψηφιακού νομοθετικού ε, συμβιβασμού, στον οποίο θα μπορούν να στηριχθούν οι πολίτες και που θα αποτελεί ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Μάλκον, τα λόγια μου αυτά τα έχω επιλέξει με πολύ προσοχή ίσως να ξεφεύγω από τα τετριμένα, από την πεπατημένη, αλλά επειδή μιλούμε για οικονομική συμφορά, χρειαζόμαστε δράση, μεγάλες δράσεις, αποφασιστικές δράσεις. Συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη οικονομική συμφορά. Ας την αναγνωρίσουμε λοιπόν, ας την παραδεχθούμε και ας αναλάβουμε τη δράση που απαιτείται επειδή ακριβώς πρόκειται για οικονομική συμφορά όρος συμβιβασμός επίσης ακούστηκε. Συμβασμός γιατί θα πρέπει για τον κάθε ένα μας να υπάρξει το δούνε προκειμένου να υπάρξει και το λαβίν. Και νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό, ότι θα πρέπει και να δώσουμε προκειμένου να λάβουμε. Θα πρέπει ο καθένας μας να κοιτάξει ένα-ένα τα κομμάτια του, μοσαϊκού και αναφέρομαι στο μοσαϊκό το οποίο αποτελεί όχι μόνο ένα συνονθήλευμα των προτιμήσεών μας ή των αλλαγών που ίσω είναι οι πιο προβεβλημένες ή οι πιο ελκυστικές, αλλά πολλές φορές οι επιλογές σε επενδύσεις έχουν εξίσου μεγάλη σημασία για τη μακροπρόθεσμη ευημερία του καταναλωτή. Στην περίπτωση της ε, περιαγωγής, αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο ε, εφόσον υπάρχει μια πραγματική ενιαία αγορά ώστε να σταματήσει να υπάρχει η επιβάρυνση περιεγωγής. Μόνο αν υπάρχει μια πραγματικά ενιαία αγορά μπορεί να πάψει να επιβαρύνεται ο καταναλωτής σε νομικούς ή οικονομικούς όρους από το κόστος της περιαγωγής και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να βάλουμε στη θέση τους ένα-ένα τα κομμάτια του μοσαϊκού. Το του θα πρέπει να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις για τις δομές. Έχω πια κουραστεί για τις, ε, να συζητάω για δομές. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ή ότι δεν πρέπει να γίνονται. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση ας το αποφύγουμε. Ας αποφύγουμε αυτές τις ε, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις γιατί και χρόνο χάνουμε και μάλιστα ο χρόνο αυτός είναι πολύ περιορισμένος. Και πρέπει να δώσουμε στον πολίτη όχι γραφειοκρατία, εν ώψη αυτής της νέας δέσμης προτάσεων και μέτρων, γιατί σε αυτό θα επιμείνω. Στον πολίτη απευθυνόμαστε και όχι στη γραφειοκρατία. Και μπορεί να χάσω κανένα δύο φίλου από, από το χώρο τη γραφειοκρατία, αλλά εγώ θα το πω και θα επιμείνω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πέραν αυτού, λοιπόν, έρχομαι με πνεύμα δεκτικό και ανοιχτό ως προς το πώς θα συγκεντρώσουμε τα κομμάτια του μοσαϊκού θα αναλάβω τις ευθύνες μου για να αντιμετωπίσω τις ε, ευθύνες και επιφυλάξει εκείνων που ανθίστανται στις αλλαγές, γιατί δεν φοβάμαι να το κάνω αυτό και η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει να φοβάμαι. Έχω αρκετή πείρα και έχω αρκετή αποφασιστικότητα. Το δυναμικό άλλωστε είναι τεράστιο. Έχω με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό αποδεθεί σε αυτόν τον αγώνα και θα σα εξηγήσω γιατί. Γιατί δεν έχει νόημα να προσπαθήσω εγώ να ταράξω τα νερά μόνη μου. Μπορεί να τα καταφέρω για μια μέρα και ένα απόγευμα να αισθανθώ ότι έχω ε, κάνει αυτό το πράγμα, αλλά αποτέλεσμα δεν φέρνω. Αλλά πρέπει να σας πω τώρα ότι έχει αλλάξει κάτι, ότι έχω υποστηρίξει από τα ανώτατα αξιώματα των θεσμικών οργάνων και με υποστηρίζουν σε αυτήν την αλλαγή πορείας, αυτή τη ριζική αλλαγή πορείας και φαντάζεστε πόσο ευγνώμων και πόσο μεγάλη τιμή αισθάνομαι όταν βλέπω ότι και αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων μου δίνουν το πράσινο φως για να προχωρήσω. όμως αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Χρειάζομαι τη δική σας υποστήριξη και είμαι πεπισμένη ότι έχουμε πολύ μεγάλο πεδίο κοινό τοποθετήσεων, μελημάτων, θέσεων, ώστε να ταράξουμε τα νερά μαζί, και το έλεγα και στον Πάλκολμ, καλά δεν θα ήταν να φέρναμε μια μικρή τρικυμία, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία στη θέση μας. Και ο πολίτης θέλει να αντιμετωπιστεί ο προβληματισμός και η ενόχληση που αντιμετωπίζει, γιατί θα το βλέπετε και εσείς στις ε, ε, εκλογικέ σα περιφέρειε ότι διαρκώ αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα ο πολίτη και σα τα εκφράζει. Περισσότερε θα είναι οι επιχειρήσει οι οποίε θα επενδύσουν εφόσον απαλληφθούν, εφόσον καταργηθούν τα τεχνητά προσκόμματα. Ε, τρίτον, οι κυβερνήσει πλέον μα λένε πρέπει να το πράξουμε. Αυτό ήταν το σαφέ μήνυμα που έχω ακούσει από παντού. Εάν λοιπόν πιστεύετε στην ενιαία αγορά, εάν πιστεύετε σε μια ισχυρή Ευρώπη, τότε μπορείτε να φέρετε αποτελέσματα που θα αλλάξουν τη ζωή του κάθε πολίτη. Και σας λέω, δεν, ας μην πιστεύουμε μόνο σε αυτή τη δυνατότητα, ας την υλοποιήσουμε. Και θα είναι η ώρα αυτή κατά την οποία θα πρέπει να σταθούμε όρθιοι και να απαντήσουμε στο προσκλητήριο και να δώσουμε την απάντηση και την ευκαιρία με αυτό το πακέτο, με αυτό τον αγώνα, με αυτό τον στόχο, στη δική σας τη θητεία και τη δική μου. Ευχαριστώ. Well, Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμότατα γιατί αφήσατε την κανονική σας ομιλία και μας δώσατε μια πολύ εμπνευσμένη ομιλία για το μέλλον της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Και ήρθατε στη σωστή επιτροπή για να, πείτε, να εκφωνήσετε αυτή την ομιλία, γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τις συγκεκριμένες προτάσεις. Πάντως ως προς το πνεύμα συμφωνούμε. Σίγουρα θα έχουμε πολλά σχόλια. Μόνο μισή ώρα μας έχει μείνει για τις ερωτήσεις. Έχω ήδη ε, γράψει αρκετούς ομιλητές. Πρώτα τον κύριο Αρίας, Εύελιν Γκέπχαρτ φυσικά, από τους σοσιαλιστές ε, η Νική Στάιλερ, Μπρος, Φανχέρν, θα ξεκινήσουμε τον κύριο Αρίας και μετά την κυρία Γκέπχαρτ. Θα ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις ε, σε δύο κατηγορίες. Πρώτο, ο Παύλο Αρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε για μία ακόμη φορά στην Επιτροπή μας να μας παρουσιάσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ψηφιακό θεματολόγιο και το πολύ φιλόδοξο και μεγαλεπίβολο σχέδιο που είχαμε γι' αυτό. Θα μιλήσω για την περιαγωγή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ιδιαίτερα με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένα θέμα που το είχαμε θίξει και στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας ε, τους, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα της περιαγωγής για τους τουρίστες ε, και τους επιχειρηματίες που κάνουν αυτό το ταξίδι από ή προς τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Εγώ θα μιλήσω για ένα καινούριο πακέτο, γιατί φαίνεται ότι το παλιό πακέτο έχει κινητοποιηθεί εξαιτία των δημοσιονομικών προοπτικών. Θέλουμε ένα backup, μία ε, λύση δευτερεύουσα αναδίπλωσης ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε τώρα γιατί θα, θα μπορέσουμε στο μέλλον να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Ε, όλοι μιλούμε για το διαδίκτυο και μάλιστα με πολύ θετικό τρόπο και όλοι πιστεύουμε στο διαδίκτυο. Όταν όμως λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις, όταν καλούμαστε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, φαίνεται ότι περνάει σε δεύτερο πλάνο το ψηφιακό θεματολόγιο και αυτό φαίνεται και από τον προϋπολογισμό. Μίζος φάρμα κατά τη γνώμη μου. Στο μέλλον ε, φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν θα επενδύσει στο ψηφιακό θεματολόγιο και στην ε, οικονομική ανάπτυξη του ψηφιακού κλάδου. Κολοσσίο λάθος κατά τη γνώμη μου. Δεν μας ενδιαφέρουν ωραίες ομιλίες, μας ενδιαφέρουν έργα για να υλοποιηθεί επιτέλους αυτή η ενιαία ψηφιακή εσωτερική αγορά. Γιατί η μεγάλη ξεχασμένη των πολιτικών των τελευταίων χρονών μάλλον είναι οι πιο νέοι. Και σίγουρα ο ψηφιακό κόσμο είναι ένα έναυσμα για να ενταχθούν και στην αγορά εργασία πολύ πιο γρήγορα. Θέλουμε να δώσουμε εναύσματα στου νέου για να ενταχθούν καλύτερα σε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Χρειαζόμαστε όμω άμεσε δράσει, ποιοτικέ και για όλου. Έχουμε ομάδα εργασία στην Επιτροπή. Μα είπατε ότι χρειάζεται τη βοήθεια όλων μα. Θα πρέπει όλοι να ανασκομποθούμε και να συσπηρωθούμε. Και ε, Είμαστε στη διάθεσή σας με την ομάδα εργασίας να σας υποστηρίξουμε και να σας ε, συνδράμουμε. Αν φυσικά είστε και εσείς πρόθυμοι για κάτι τέτοιο για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και ανάλυση των δυνατοτήτων για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Φυσικά θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτό το πακέτο που μας ε, αναγγείλετε. Ε, θα σας στείλουμε χειροβοηθίες. Είμαστε πρόθυμοι, όπως είπα, να σας συνδράμουμε και ό,τι μελήσουμε να κάνουμε τώρα, πολύ γρήγορα θα καλύψουμε στο μέλλον ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει πρώτα να εξυπηρετεί τους πολίτες μας που είναι πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι και φυσικά να εξυπηρετεί και τις επιχειρήσεις μας. Το ψηφιακό θεματολόγιο μέχρι τώρα έχει τροποποιήσει, ευνοήσει τις, ε, τα εθνικά ψηφιακά θεματολόγια όπως το ισπανικό που προώθησε ο Υπουργό Σόρια. Ερωτώ λοιπόν, το νέο πακέτο που μας αναγγείλατε ποιες αλλαγές θα επιφέρει στην, ε, στις εθνικές προτάσεις και στις εθνικές καταστάσεις. Ε, θα γίνει μια, ένα βήμα προς τα μπρος ή θα υπάρξει μια παλινδρόμηση με το νέο πακέτο. Η Εύελιν Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κυρία Κρούς για το φρέσκο πνεύμα με το οποίο μας ε, κάνατε την, την παρέμβαση, την ομιλία. Μιλήσατε και ως πολιτικός πρέπει να πω, πράγμα το οποίο Ιδιαίτερα με ευχαρίστησε, που προς τώρα πολιτικός και όχι ως θεωρητικός. Πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε τότε. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να δίνουμε στον πολίτη ε, παρουσιάσεις και θεματολόγια περιορισμένα και τεχνικού χαρακτήρα για περιορισμένο αντικείμενο. Πρέπει να του δώσουμε μεγάλες προοπτικές και λύσεις. Το υπογραμμίσατε κι εσείς στους νέους ιδιαίτερους θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση, γιατί αυτή είναι το μέλλον και για αυτούς άλλωστε φτιάχνουμε και την νομοθεσία. Εμείς το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας το έχουμε πια διανύσει. Οι νέοι σήμερα έχουν άλλη, άλλη συμπεριφορά και στάση στην κοινωνία, διαφορετική από τη δική μας. Όταν ήμασταν εμείς νέοι δεν είχαμε αυτές τις ε, τεχνολογικές δυνατότητες και έτσι αυτοί οι νέοι δεν χρειάζονται σχεδόν ούτε καν τηλεόραση στο σπίτι να έχουν, γιατί έχουν τον υπολογιστή τους και μπορούμε τον υπολογιστή να δουν οτιδήποτε, οποιοδήποτε περιεχόμενο τους ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν αυτή τη νέα ψηφιακή κοινωνία πρέπει να την περιγράψουμε και να την λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αναφέρατε πολύ σημαντικά θέματα. Καταρχάς το θέμα της περιαγωγής, το θίξατε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και να πληρώνουμε τέλος περιαγωγής. Δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται και γι' αυτό έχετε την πλήρη υποστήριξή μου, την πλήρη υποστήριξη της ομάδας των Σαρδημοκρατών στον αγώνα της ε, αντιμετώπισης αυτών των τελών περιαγωγής. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όταν ταξιδεύω μεταξύ του ΚΕΛ και του Στρασβούργου, που έχουν πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, να πληρώνω περιαγωγή και δεν πληρώνω περιαγωγή όταν ταξιδεύω από το ΚΕΛ στο Βερολίνο, που χωρίζουν πάνω από χίλια χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για τους νέους, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα. Η ουδετερότητα του δικτύου είναι το α και το ω όλες τις υπόθεσεις νομίζω, η ουδετερότητα του δικτύου. Βλέπω στη Γερμανία, επί παραδείγματι, μια μεγάλη εταιρεία η οποία ε, προσπαθεί να ξεφύγει από την υποχρέωση της ιδιωτερότητα του δικτύου. Αυτό με κάνει να καταλήξω στο συμπεράσμα ότι οπωσδήποτε χρειάζεται η ιδιωτερότητα του δικτύου και δεν είναι δυνατόν με μονομένε εταιρείε όπω συμβαίνει στη Γερμανία να μα λένε ότι α, κοιτάξτε, θα πρέπει να αυξήσουμε το κόστο τη πρόσβαση ή να καθυστερούμε αντίστροφα την, λειτουργία του δικτύου, να είναι πιο βραδία δηλαδή ε, η λειτουργία του δικτύου, εάν έχετε μεγάλη πρόσβαση, για πολλή ώρα πρόσβαση σε πολλά γιγαμπάιτ πρόσβαση στο δίκτυο. Δεν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή όπου έχουμε τη χρήση του δικτύου για τα πάντα, για τηλεόραση, για παιχνίδια, για μουσική, για όλα, να ε, επιβραδύνεται ή να κοστίζει περισσότερο η χρήση, η ποσότητα του, ε, της χρήσης του διαδικτύου. Πρέπει να έχουμε διαφορετικές μεθόδους και χρήσεως και πληρωμής ή επιβάρυνσης που θα πρέπει να εξεταστούν και θα πρέπει να φροντίσουμε ακόμη και εκείνος ο οποίος δεν έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν είναι δυνατόν, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, να αυξάνονται ραγδαία ε, οι τιμές πρόσβασης στο διαδίκτυο, τα τέλη ε, χρήση διαδικτύου. Γι' αυτό λοιπόν σας υποστηρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια στο να εξασφαλίσετε για όλους τους πολίτες την πρόσβαση και τη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θέλετε να ακούσουμε και ακόμη μια ερώτηση και να απαντήσουμε, κυρία Στάιλερ. Θα συνδέσουμε. Εκτός αν θέλετε να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις πρώτα και μετά να απαντήσετε συνολικά. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την καταπληκτική της ομιλία. Μιλήσατε για τους νέους, ε, για τους ε, πιο ηλικιωμένους, αναφερθήκατε στην υγεία και τη μοναξιά στη... όταν κανείς είναι πιο ηλικιωμένος. Και η μαμά μου πήρε το πρώτο της smartphone και πήγε στην εκκλησία. Ε, ε, και πραγματικά ε, ήταν κάτι καινούριο για αυτή το άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες. Ε, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι κάνουν αυτό το άνοιγμα προς την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι μια επιπλέον πρόκληση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αρκετή πρόσβαση και στις βιβλιοθήκες και θέλουμε περισσότερο δημόσιο χώρο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσκοπτη σύνδεση Πολύ σωστά είπε η Εύελιν ότι έχουμε αυτό το ψηφιακό μέρισμα και την κοινωνική ένταξη, αλλά είναι και το θέμα της γνώσης. Θα πρέπει αυτή την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε και να μην στερήσουμε τη γνώση στους νέους, την ανοιχτή πρόσβαση. Για μας μπορεί να ήταν κάτι δεδομένο, αλλά για τους νέους θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για να εξασφαλίσουμε αυτή την ανοιχτή και εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στη σύνδεση. Σας ευχαριστώ και μας άρεσαν τα tweets που μας στείλετε. Έχουμε και εμείς στην Επιτροπή tweets και είμαστε και στο Twitter. Θα πρέπει και στο σημείο αυτό να ενεργοποιηθούμε και έχετε απόλυτα δίκιο. Φαντάζομαι το, θα στείλετε με tweet ε, την ομιλία της κυρίας Κρούς. Φαντάζομαι το έχετε φροντίσει ήδη. Η Ρόζα Τιν. Μετά ο κύριος Μάντερς. Ο καθηγητής Κορέρα δηλαδή, Κάμπος, τον ξέχασα. Και η κυρία Μπέλα επίσης. Να επαναλάβω τη σειρά. Κορέα Δε Κάμπος, μετά η Ροζατίν, Χέρν, Μάντερς και μετά η κυρία Μπέλα. Ξέχασα το μικρό σας όνομα, αλλά θα το μάθω που θα μου πάει. Αντώνιο Κορέντε Κάμπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας και να σας συγχαρώ για το ότι αναγνωρίσατε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε έναν οικονομικό όλεθρο και αναγνωρίσατε ότι η ανεργία των ε, νέων είναι ίσως ε, το πιο σοβαρό μας πρόβλημα. Και είπατε ότι ελπίζετε το ψηφιακό θεματολόγιο να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης. Σας ευχαριστούμε για αυτά γιατί πρόκειται για μια αναγνώριση έστω και, και καθυστερημένη της σοβαρότητας της κατάστασης και είναι πολύ χρήσιμη αυτή η αναγνώριση. Θα σας παραθέσω μια εμπειρία που είναι πολύ οικία πια το τελευταίο καιρό. Στις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, εκεί που το τραπεζικό σύστημα χωλαίνει και είναι σχεδόν ανύπαρκτο το τραπεζικό δίκτυο, αυτό δεν έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές αυτό, αλλά χρησιμοποιούν τα κινητά τους ως υποκατάστατο για τις εμπορικές τους συναλλαγές. Γιατί μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορούν να κάνουν αγορές και ουσιαστικά μπορούν ακόμη και να εκδίδουν επιταγές ή και να ε, πληρώνουν απλές ε, εμπορικές συναλλαγές. Φαίνεται ότι η χρήση του κινητού για, για τέτοιου είδους δραστηριότητες έχει τεράστια άνθηση και στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Φαίνεται ότι οι καταναλωτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο ψηφιακό σύστημα από τις τράπεζες. Προτιμούν το ψηφιακό σύστημα γιατί το τραπεζικό σύστημα δεν αξίζει εμπιστοσύνη κατά τη γνώμη τους. Και αυτή η ιδέα της εμπιστοσύνης και η αρχή της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντική. Και έρχομαι εδώ στην ε, βασική μου ερώτηση. Είπατε ότι τα σύνορα δεν έχουν λόγο σε μια ψηφιακή οικονομία. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Μια ψηφιακή οικονομία δεν πρέπει να γνωρίζει σύνορα και όρια. Δεν έχει νόημα να έχουμε ε, αυτά τα τεράστια, αυτούς τους τεράστιους φραγμούς ε, των τιμών και τα υπέρογκα τέλη του roaming, της περιαγωγής. Είχαμε πολύ άριθμες συζητήσεις ε, και με δικούς υπαλλήλους στην Επιτροπή και η το επιχείρημα που μας έδωσαν για τις τεράστιες διαφορές των τιμών είναι ότι θέλουμε να αφήσουμε την τιμή, την ε, αγορά να ανθίσει, να εμφανιστούν νέοι ε, φορείς, νέοι operators, αλλά τελικά δεν δημιουργήθηκαν, ε, δεν είχαμε πολύ περισσότερους φορείς στην αγορά, πολύ περισσότερους operators. Και μπορεί να έχει μειωθεί η τιμή, αλλά ελάχιστα η περιαγωγή εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, πολύ δαπανηρή. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτό το θέμα για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό σύστημα. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία να αρχίσουμε επιτέλους ε, να σκεφτόμαστε ποια θα είναι το καλύτερο ανώτατο όριο, το καλύτερο πλαφόν για την περιαγωγή. Ευχαριστώ κυρία Τιούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάλκολ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την ομιλία της. Λυπάμαι γιατί έφτασα κάπως καθυστερημένα, γιατί όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς έκλεισαν τα τούνελ στις Βρυξέλλες και αυτό και έμεινα μπλοκαρισμένη στη συμφόρηση. Εν περιπτώσει δεν είναι δικαιολογία αυτό, αλλά καθυστέρησα έτσι. Συμφωνώ με την Εύελιν ότι η ομιλία σας έχει μείζωνα πολιτική σημασία γιατί η πολιτική στην Ευρώπη θα πρέπει να άρει τα όρια και τους φραγμούς της εσωτερικής αγοράς, τα σύνορα που ουσιαστικά χωρίζουν τους πολίτες. Και σίγουρα από αυτήν την άποψη η περιαγωγή είναι από τα πιο νευραλγικά σημεία αυτών των ορίων και των φραγμών. Ζητήσατε να συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια ανάληψη κοινών δράσεων και συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ και με τους συναδέλφους ότι χαιρόμαστε για την προσήλωσή σας στο θέμα αυτό και την ε, μεγάλη στράτευση που δείχνετε, γιατί πραγματικά αυτό θα είναι βασικό ε, σημείο που διχάζει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και ε, χαίρομαι για τον ενθουσιασμό που δείξατε για μια μεγαλύτερη και βαθύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χάρη και στο ψηφιακό τομέα. Συμφωνώ με αυτά που λένε οι συνάδελφοι και εσείς ότι δεν έχουν νόημα τα όρια, δεν έχουν όριμα τα σύνορα. Και τώρα για την ε, ε, online επίλυση των διαφορών, για την ε, επίλυση των διαφορών μέσω διαδικτύου θα επιλύσουμε καλύτερα τα προβλήματα και των καταναλωτών και ε, των, των διαφόρων επιχειρήσεων και μάλιστα μπορεί να γίνεται αυτό σε όλες τις επίσημες γλώσσες, κάτι που θα δώσει μεγάλη αίσθηση ασφάλειας και στις επιχειρήσεις και σε, στους καταναλωτές. Γιατί και εκεί έχουμε έναν φραγμό που θα πρέπει να άρουμε. Υπάρχει όμως ένα οικονομικό πρόβλημα και το γνωρίζουμε. Και αυτή είναι η ερώτησή μου το, το θέμα της ε, online επίλυσης των διαφορών, της επιγραμμικής επίλυσης των διαφορών θα το συμπεριλάβετε στις προτεραιότητές σας και στα προγράμματα που θα, χρηματοδοτούν, θα χρηματοδοτηθούν, ελπίζω, από το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη, από το Connecting Europe Facility. Είναι προφανές ότι είναι ένα από τα στοιχεία του ψηφιακού θεματολογίου και θα είναι και ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του ψηφιακού θεματολογίου Πιστεύω ότι έτσι θα ενισχύσουμε τις ε, δράσεις και την ε, ψηφιακή αγορά που σας είναι τόσο προσφυλής και σε εμάς το ίδιο. Και ελπίζω να βρούμε κονδύλια για κάτι τέτοιο. Γιατί είναι κοινή μας υποχρέωση και δική σας και δική μας, κοινή μας υποχρέωση και καθήκον απέναντι στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Ακρούς να μας ε, μιλήσετε για αυτή την εμπνευσμένη ομιλία. Βλέπω ότι προσπαθείτε με όλες σας τις δυνάμεις να αντιμετωπίσετε το θέμα των τελών περιεγωγής, γιατί είναι όντως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Από αυτό θα εξαρτηθεί και πολύ η αποδοχή, αλλά και πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Πάντα βέβαια έρχονται οι επιχειρήσεις και λένε θέλουμε πιο πολλά χρήματα, χρειάζομαστε υποστήριξη για να μπορέσουμε να επενδύσουμε, για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να έχουμε νέα μέσα αναχρηματοδότησης από τις ε, συμβάσεις με τον ε, πελάτη. Αυτό το βλέπουμε και στο ε, roaming, την περιαγωγή, αλλά και σε άλλα θέματα που όμως αποτελούν τελικά μεγάλο πρόσκομα και φραγμό στην εξελίξη του τομέα αυτό. Ε, ιδιαίτερα όμως εμένα με ενδιαφέρει το θέμα της ουτερότητας ε, του δικτύου, το έθιξε η κυρία Γκέπχαρτ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δική μου γνωμοδότηση επεξεργασία για το ε, νέφος, για το ψηφιακό νέφος και ένα ζήτημα που έχουμε να κάνουμε, με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι η αξιοποίηση του νέφους και η δυνατότητα να μην επιλέγει ο ίδιος ο πάροχος της των υπηρεσιών, την ποιότητα ή την ταχύτητα ή τον όγκο των πληροφοριών που μπορούμε να ε, θέσουμε σε κυκλοφορία μέσω του νέφους, του ψηφιακού νέφους, αλλά να μπορεί ο πελάτης ο ίδιος να το επιλέγει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα θέματα να εργαστούμε κατά τρόπο διαρθρωμένο, χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση ευρωπαϊκό δίκαιο η, η οποία θα διασφαλίζει την ουτερότητα του δικτύου, γιατί πάντα θα δούμε επιθέσεις όπως είδαμε πρόσφατα στη Γερμανία που ε, εις βάρος της του δικτύου και όπου θα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι ε, πριν, μπορούμε να έχουμε ένα πάγιο τέλος το οποίο δεν θα μπορεί να ε, ανεβαίνει περαιτέρω ή αλλιώ, αν κάποιο θέλει ένα φθηνό πακέτο, τότε μπορεί να έχει μια επιπλέον επιβάρυνση σε περίπτωση που ξεπεράσει το πακέτο του. Αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένα πάγιο τέλο το οποίο δεν θα αυξάνεται σε καμία περίπτωση. Και όλα αυτά πάντα σε ε, σχέσεις διαφάνειας ως προς το κόστος για τον πελάτη. Πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης, ο χρήστης του δικτύου, ε, τι πληρώνει και γιατί το πληρώνει. Ε, είναι πολλές οι συνθάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενημέρωση ικανοποιητική και βλέπουμε ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν είναι ικανοποιητικές οι συνθήκες πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου που προσφέρουν κάποιες από αυτές τις συμβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν και νομίζω ότι εκπροσωπώ όλη την Επιτροπή όταν, λέγοντας, όταν λέγω ότι το, ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και πρέπει να το αξιοποιήσουμε για μια πραγματική ψηφιακή εσωτερική αγορά για την Ευρώπη που χρειαζόμαστε, κάτε επιγόντως και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, με υποστήριξη και για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεν είναι σε θέση αυτόνομα να ε, δραστηριοποιηθούν και αν δεν θέλουμε να χάσουμε το μεγάλο δυναμικό που έχουν ορισμένε περιοχές της υπαίθρου για ανάπτυξη ε, επιχειρησιακή, επαγγελματική, τότε θα πρέπει να λύσουμε ακριβώς το θέμα του νέφους ε, και της ψηφιακής διασυνδεσιμότητας και του εργοστηρικίου. Ευχαριστώ πολύ. Μάντερ, Σαμπέλ. Και μετά τη Είναι τελευταίοι σχεδόν θα εξαντλήσουμε το χρόνο μας. Βέβαια ξεκινήσαμε λίγο αργότερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Μπορούμε να παρατείνουμε λίγο το χρόνο. Κυρία Κρούς, έχω δύο ερωτήσεις. Είστε πολιτικός με όραμα και με πολύ σύγχρονη σκέψη. Και πραγματικά ελπίζω να ανανεωθεί η εντολή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τέτοιους επιτρόπους χρειαζόμαστε. Ε, ε, επιτεθήκατε και στη Microsoft και σε μεγάλους γίγαντες ε, του ψηφιακού κόσμου για να βελτιώσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις τηλεπικοινωνίες σας. Η, σας υποστηρίζουμε λοιπόν. Ακόμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε παμπάλαιους υπολογιστές, ακόμη έχουμε Microsoft προγράμματα του 2003 θα πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα βήμα προς το σύγχρονο κόσμο. Πιστεύω ότι με το δικό σας δυναμισμό θα δώσετε δυναμισμό και θα εξυγχρονίσετε και τα θεσμικά όργανα. Γιατί ε, καλό θα ήταν να εξυγχρονιστεί και η Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Και αν είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ κυρία Σαμπέλα. Αμπέλα. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Φυσικά, πολλά σημαντικά ακούστηκαν στην ομιλία σας. Πολλά συνδέονται και με την ε, κοινωνική ατζέντα, με το κοινωνικό θεματολόγιο. Μεταξύ αυτών, είπατε ότι εμείς θέλετε να πάμε στους εκλογείς μας και να τους πούμε ότι θα μειώσουμε το κόστος της Αυτό φυσικά είναι καλό για τους καταναλωτές, γιατί θα υποφεληθούν από μια τέτοια κατάσταση. Και το άλλο που είπατε αφορά τη νέα γενιά και την ανεργία των νέων. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Οι καταναλωτές θα πρέπει να υποφεληθούν από το τέλος, την πάυση του τέλους της περιαγωγής, αλλά οι εταιρείε θα πρέπει να επενδύσουν για να Προσφέρω περισσότερες θέσεις εργασίας στους νέους για να μειωθεί η ανεργία τους. Συμφωνώ απόλυτα με την πάυση του τέλους περιαγωγής. Πώς θα γίνει αυτό και πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων, θα ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Uh, Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τσασκόφσκι, θα ήθελα όλοι να σοπάσετε, γιατί είναι δύσκολο να ακούσουμε τους ομιλητές. Παρακαλώ, ε, φωνασκείτε εκεί πίσω στα έδρανα των πολιτικών συμβούλων. Κύριε Τσασκόφσκι, έχετε το λόγο. Θέλω να μιλήσω για την προσπελασιμότητα του ίντερνετ είναι ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς. Ε, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά τους μεγαλύτερους στην ηλικία και θα πρέπει να αλλάξουμε την, τον τρόπο προσέγγισης ε, από τις διακρίσεις να πάμε στην πρόσβαση για όλους. Συγχαίρω την Κομισιόν που το πρότεινε, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία. Θα ήθελα να με στηρίξετε. Γιατί ως προϋπόθεση προτείνεται να αντιμετωπίσουμε μόνο ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη δέσμη υπηρεσιών με αυτή την υπηρεσία. Όχι, θα πρέπει ε, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να προσπελάβνονται ε, χωρίς προϋποθέσεις. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα. Λίγο πιο μεγάλη φιλοδοξία, γιατί είναι από τους τομείς της αγοράς που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της γενικά στην ε, ενιαία αγορά. Η κυρία Ρέντινγκ, λέει ο Μάλκομ, θα απαντήσει. Ω, συγγνώμη, την κυρία Κρούς εννοούσα. I Πω, πω, αμηχανία. Ε, αυτό δείχνει πόσο πολύ έχω κάτσει σε αυτή την καρέκλα. Μπερδεύτηκα. Επιτρέψτε στην κυρία Ρέντινγκ πάλι να σας απαντήσει, εξασφαλίζοντάς της όμως την ησυχία στην ε, αίθουσα. Θα γράψω το όνομά μου, λέει η κυρία Κρούς, σε ένα χαρτί για να το έχει μπροστά του Μάλκομ. με απευθύνουν με διαφορετικούς τρόπους. Ε, εξηγείται από το γεγονός ότι έχω κάνει και πολλούς γάμους. Έχω πολλούς γάμους στο ενεργητικό μου. Δεν θα αναφέρω τα ονόματα των ευρωβουλευτών που μίλησαν για να εξοικονομήσω χρόνο και αν δεν σας απαντήσω τώρα, θα σας απαντήσω γραπτός αργότερα. Ούτως ή άλλως ε, η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και σε σερβίρουμε και καφέ. Αυτά που είπατε για τη μητέρα σας ε, με συγκίνησαν. Γιατί καμιά φορά ρωτάω, πού βρίσκεται την έμπνευσή ε, σας. Με ρωτάνε μάλλον πού βρίσκω την έμπνευσή μου. Την πρώτη α, εβδομάδα που ήμουν στο γραφείο, ήμουνα σε ένα γεγονός όπου υπήρχαν νέοι ε, επιχειρηματίες, εφευρέτες κτλ. Δίπλα μου καθόταν κάποιος που μιλούσε για την έμπνευσή του σε κάποιον άλλον. Και του λέω, μιλάς αυτό στο, στον ανταγωνιστή σου μου λέει «Είσαστε πολύ παλαιομοδίτης, Επίτροπε». Δεν έχετε καταλάβει ότι πρέπει να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε. Είναι ε, ένα μάθημα που διδάχτηκα, κάτι που έμαθα εκείνη τη μέρα. Η γενιά μου κρατούσε τα κεκτημένα της και προσπαθούσε να κάνει δουλειές, να αυξήσει τα κέρδη. Και αυτός μου είπε ότι τα αποτελέσματα που θα έχω είναι καλύτερα αν ακούσω και μοιραστώ. Η άλλη μου έμπνευση είναι η εγγονή μου. Ε, είναι Αμερικανή, μένει στο Σαν Φρανσίσκο, είναι πεντάχρονη και επικοινωνούμε το, τα Σαββατοκύριακα. Κάποια στιγμή μου λέει «Α, δεν σε εννοούμαστε γιαγιά». πεντάχρονο μου το είπε αυτό. Της λέω «Ορίστε». Μου λέει «Εγώ έχω τις δικές μου αρχές και εσύ έχεις τις δικές σου». Τη λέω, μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Και μου λέει, όχι, είσαι πολύ γριά γι' αυτό. Και σκέφτηκα λοιπόν, όχι, θα αποδείξω ότι δεν είμαι τόσο μεγάλη. Αυτές τις εμπνεύσεις τις πήρα από την πεντάχρονη γονή μου και από εκείνον τον εφευρέτη που ήταν 14 χρονών. Ένα άλλο θέμα που θίξατε όλοι σας είναι η ενεργεία των νέων. Δεν είναι μόνο εφιάλτη σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε με αξιοπρεπή τρόπο αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φρικόδεις ε, συνέπειες. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν ποτέ να παντρευτούν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να βρουν διαμέρισμα, να μείνουν μόνοι τους, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει προοπτική. Και ξέρω πολύ καλά ότι στην ψηφιακή οικονομία υπάρχει τρόπος, ε, είναι αυτό ένα εργαλείο για να αλλάξουμε την οικονομία μας. Και ούτω ή άλλως ε, με την ψηφιακή αυτή οικονομία συνδέεται πολύ περισσότερο η νέα γενιά. Αυτή η μεγάλη ε, συμμαχία, ο συνασπισμό, μεταξύ οργάνων και επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός, ούτω ώστε να πάμε online, να δούμε, να δώσουμε το βιογραφικό μας, να δούμε τι προσόντα έχουμε, ε, πού μπορούμε να βρούμε δουλειά κτλ. Και επίσης μην ε, υπονο, ε, υποτιμάτε την, ε, τις νέες επιχειρήσεις. Δεν, είναι παντού στην Ευρώπη, όχι μόνο σε ένα-δυο κράτη-μέλη, οι νέες επιχειρήσεις. Επομένως, όταν θέλουμε να μιλήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την ε, ανεργία των νέων, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μέσω της ψηφιακής οικονομίας. Και μην ξεχνάμε εδώ και τι γυναίκε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στι δύσκολε εποχέ τις ξεχνάμε τις γυναίκες. Η θέση μου είναι ίση μεταχείριση. Αυτή είναι η απάντηση που δίνω. Επίσης όλοι μιλήσατε για την περιαγωγή. Και το είπα κι εγώ. Κοιτάξτε, μιλάμε για φοβερά δημοφιλές θέμα, έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά είναι μία ψηφίδα σε ένα πάζλ. Και εγώ θα το εξασφαλίσω αυτό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κομμάτι από το παζλ χωρίς τα υπόλοιπα. Αυτό το παζλ θα λειτουργήσει χάρη στην εμπλοκή σας, χάρη στη θέλησή σας να προχωρήσουμε μαζί. Ehm, Όταν ταξιδεύει κανείς στο εξωτερικό, στην Άπο Ανατολή, στην Εθνική Αμερική, όλοι μας λένε τι τυχεροί που είστε που έχετε την ενιαία αγορά, τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του κόσμου. Αλλά πώς τη χρησιμοποιείτε? Και αυτό είναι το ερώτημα εδώ. Τι την κάνουμε? Όλα συνδέονται με τον ανταγωνισμό. Ένα-δυο από εσά ε, είπατε Τελικά, ποια είναι η επίπτωση στην αγορά όλων αυτών. Εγώ πιστεύω πολύ στον ανταγωνισμό. Γιατί. Γιατί δίνει τις εγγυήσει στον καταναλωτή για ισότιμη, ισότιμο παιχνίδι όλων των παιχτών στην αγορά, ε, εξασφαλίζει την καινοτομία, γιατί αν δεν πιέσουμε για καινοτομία, χάνουμε και θα χάσουμε το οποιοδήποτε πλεονέκτημα έχουμε απέναντι στους ε, ανταγωνιστές μας. Το θέμα δεν είναι να περιχαρακώσουμε την Ευρώπη. Εδώ πέρα έχουμε ένα παγκόσμιο κόσμο. Επίσης, πολλοί από εσά αναφέρατε την ε, εμπιστοσύνη. Τη λέξη εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Ε, εντυπωσιακή λέξη. Να σας πω κάτι. Τι ανακαλύψαμε. Υπάρχει και στην επισκόπηση του ψηφιακού θεματολογίου ούτως ή άλλως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αλλά δεν είναι το μόνο, ούτε το χειρότερο. Η Ιταλία. Μια ανοιχτή, δημοκρατική χώρα. Στην Ιταλία, το 41% των Ιταλών δεν έχουν ποτέ ε, μπει στο ίντερνετ. Γιατί? Εντυπωσιακό. Σε άλλα κράτη-μέλη Και δεν είναι μεμονωμένο παράδειγμα η Ιταλία, έτσι. Ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ίσως. Και, και κυρία Στάιλε, δεν είναι όλοι σαν τη μαμά σας. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα που πολλοί δεν μπαίνουν στο ίντερνετ, το θέμα της εμπιστοσύνης. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι παίζει και εμπιστοσύνη εδώ. Δεν ξεχνάτε ότι σε άλλες υπήρους έχουν γίνει τρομερά βήματα. Η Αφρική είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ενδιαφέρουσα είναι και η θέση των γυναικών χάρη στα κινητά τηλέφωνα, χάρη στη δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών, μικροπιστώσεων, μέσω των κινητών, μέσω της κινητής τηλεφωνίας. Χάρη σε αυτό είναι πιο ανεξάρτητη μπορεί να ξεκινήσουν νωρίτερα την, επιχείρηση, την επιχείρησή τους και είναι πολύ πιο ασφαλές να κινείσαι χωρίς λεφτά στην τσέπη σου βέβαια, αλλά με ψηφιακό χρήμα. Επίσης, όλα αυτά που λέω είναι ένα πακέτο. Τι κάνουμε, επανέρχομαι στην ανεργία των νέων. Η ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντική. Γιατί αν η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα, γιατί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, αυτό σημαίνει ότι και ο ανταγωνισμός θα παίξει το ρόλο του. Αυτό συνδέεται όμως και με την εκπαίδευση, συνδέεται με τις δεξιότητες. Γιατί ένα άλλο θέμα, Μάλκομ, και το ξέρουμε και δεν είναι περίπλοκο να το σκεφτούμε, είναι ότι μέχρι το 2015 θα χρειαστούμε ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης να καλυφθούν, ε, που συνδέονται με την κοινωνία των πληροφοριών. Είναι πρόκληση αυτό. Ε, όχι μόνο να εξασφαλίσουμε δουλειά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά να βάλουμε σε αυτές τις θέσεις ανθρώπους, ούτως ώστε να μην αναγκάσουμε τις εταιρείες να στραφούν αλλού για να βρουν τα, τα εργατικά χέρια που χρειάζονται. Να τους τα δώσουμε εμείς. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, πώς μπορούμε να συνδέσουμε τις τεχνικές ανάγκες με τις δεξιότητες κτλ. Καμιά φορά εδώ μπαίνει και το θέμα της α, κινητικότητας. Δεν μπορείς να δεις τους φίλους σου γιατί είναι μακριά ας πούμε. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, βεβαίως από τη μία, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ψηφιακές ευκαιρίες δίνουν την απάντηση. Παραδείγματος χάρη, ο ερευνητής μπορεί να έρθει σε επαφή με μία επιχείρηση χωρίς να είναι στο ίδιο μέρος. Μία γερμανική εταιρεία, ας πούμε, ξεκινάει ένα κέντρο στην Ισπανία. γιατί ξέρει ότι τα προσόντα που έχει ανάγκη βρίσκονται εκεί. Κινητικότητα λοιπόν είναι η απάντηση. Πόσο χρόνο έχω, καθόλου, ο Μάλκομ. Να μιλήσω για την ουδετερότητα του δικτύου. Ξέρετε τις δεσμεύσεις μου. Μην, το ξεχνάτε. Το έχω πει και το ξαναλέω. Ανοιχτός και απρόσωπος χαρακτήρα στο δίκτυο. Αυτό για μένα είναι θέσφατο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα τα εμπόδια παρεμποδίζουν τον, τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι απαράδεκτο, το λέω ξεκάθαρα. Θα δω όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας και θα τις απαντήσω γραπτός. Μπορείτε να μας στείλετε email, ψηφιακή απάντηση εξάλλου. Σας ευχαριστούμε. Είδατε πόσο θερμά σας χειροκρότησαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε Κρούς, αυτή τη φορά. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, ούτως ώστε και να ταράξουμε τα νερά και να βάλουμε το πλοίο, να το φέρουμε πίσω στο λιμάνι, harbor, όπως το όνομα του Προεδρού αστείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ας κάνουμε σήμερα ε, την απαρχή του κινήματος της 30ης Μαΐου. Ας είναι αυτή η μέρα που θα γιορτάσουμε αυτό το κίνημα. Η 30η Μαΐου. Um, Ευχαριστώ συνάδελφοι που μας δώσατε λίγο χρόνο. Νομίζω ήταν καλή η ανταλλαγή απόψεων για μείζωνα πολιτικά θέματα με την Επίτροπο. Αντίγραφα του, της ομιλίας της κυρίας Κρούς θα σας δοθούν και όλα όσα σας υποσχέθηκε θα, τα, θα σας τα δώσει. Λοιπόν, το πρώτο σημείο α, στον κατάλογο ψηφοφορίας είναι το υπολογιστικό νέφος. Κυρία um, κυρίας Βαν Χέιεν, που είναι, δεν είναι, ας ξεκινήσουμε χωρίς αυτήν. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Πολύ θέλετε να ξεκινήσουμε. Αδειμονείτε. Πάραφος 1. Τροπολογία 15. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 32 είναι εδώ. 29 κάρτες έχουμε από ό,τι φαίνεται. 31 ανεβαίνει το νούμερο. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι, δεν περνάει. 18 κατά, 13 υπέρ. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 16 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά απορρίπτεται 29 υπέρ κατά απορρίπτεται ε, τροπολογία 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 50 υπέρ κατά εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 57 υπέρ. Υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 κατά, 16 υπέρ. 58 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Πολύ κοντά είναι τα δύο στρατόπεδα. Ψηφίσουμε ξανά την 61 ηλεκτρονικά. Γρήγορα παρακαλώ. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 16 κατά. 62 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Οι αναφορές. On μπλοκ Από 1 έως 5. Υπέρ, κατά εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις, ε, τροπολογία 6, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 8, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 13, υπέρ, κατά, εγκρίνεται προφορική τροπολογία στο, στην αιτιολογική σκέψη υπέρ κατά γκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τελική γνωμοδότηση. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 33 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά. ευχαριστώ κυρία Φερχέιν και ελπίζω να πάτε στην Επιτροπή Βιομηχανίας και να υποστηρίξετε την γνωμοδότησή μας, γιατί για αυτή την κάναμε. Και τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Φόξ. Κατσαν. Για τυχερά παιχνίδια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες μέχρι αργά το βράδυ για τις συμβαστικέ τροπολογίες. Έχουμε μία προσαρμογή που θα την ακούσετε μετά. Ο εισηγητή θα ήθελα παρακαλώ να πει δυο λόγια. Άσλι, η κυρία Πιετικάινεν πάντως θέλει να κάνει μία δήλωση. Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το αφοσιωμένο έργο τους. Είναι μια καλή συμβαστική λύση πιστεύω και ευχαριστώ ιδιαίτερα και το προσωπικό μας τους βοηθούς από τις πολιτικές ομάδες. Ξέρω ότι έχουν δουλέψει και περασμένα μεσάνυχτα ακόμα για να φτάσει αυτή η δουλειά στα τραπέζια μας. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια ιδιαίτερα την Ντάινα, τη δική μου βοηθό σε ένα τεχνικό ζήτημα τώρα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει όλες τις συμβαστικές ε, προτάσεις και ότι δεν αναφέρεται το, ο τίτλος της πολιτικής μας ομάδας για τεχνικούς λόγους μαζί με, τους, ε, με τις συμβαστικές προτάσεις. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα λοιπόν ε, αυτό για το οποίο αποσύρει την 48, 51, 2, 2, 3, 309, 368 Ξέρω ότι δεν προλάβατε να τις γράψετε, αλλά δεν πειράζει. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προλαφθεί για, για το τελικό κατάλογο ψηφοριών. Ευχαριστώ. Στην συμβαστική 8 παρακαλώ να ρίξετε μια ματιά γιατί έχουμε διαφορές, έχουμε αποκλήσει ως προς τις προφορίες. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Πολύ καλά λοιπόν ομού της 84 έως 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 89 υπέρ κατά εγκρίνονται συμβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 116-119 μαζί. Παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται. Mm Και 120 πήγαινε μαζί με τις προηγούμενες τροπολογίες, άρα περνάμε στην 126, 127, 128, τρεις τροπολογίες μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. 126, 127, 128. Πέρασε τη προφορίες. Απερίφθησαν. Απερίφθη η διαγραφή δηλαδή. Συμβαστική 8. Σε τμήματα. Για να είναι σαφή η κατάσταση, το βλέπετε στον κατάλογό σα, αλλά με λάθο σειρά βλέπετε τα τμήματα. Δηλαδή η πρώτη τμηματική ψηφοφορία, απλά η 8 χωρίς τις λέξεις τμήμα 2, τμήμα 3, part 2, part 3. Είναι αυτό που βλέπετε πρώτο στη σειρά. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται λοιπόν. Το δεύτερο κομμάτι τώρα είναι το τρίτο που βλέπετε και όχι το δεύτερο. Α, όχι, το αλλάξατε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε το πραγματικό δεύτερο κομμάτι. Takes note of the Commission's work on the infringement cases. Λαμβάνει υπόψη τη δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις παραβιάσεων κτλ. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Υπέρ, όπως το βλέπετε στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Να το ξαναδιαβάσω, το takes part, takes note of the commission's work. Λαμβάνει υπόψη τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υποθέσεις παραβάσεως κτλ. Ξεκινάει η ψηφοφορία για το κομμάτι 2, όπως το βλέπετε στον κατάλογο των ψηφοφοριών και όπως σας το διάβασα. Λίγο πιο γρήγορα σας παρακαλώ να ψηφίζετε. Γιατί ξέρετε με τα ηλεκτρονικά καθυστερούμε. πέρα εγκρίνεται. Ο κύριος Άστον. Φόξ. Πρόεδρε, εγώ νόμιζα ότι το 3 είχε εγκαταληφθεί. Το some of which have been dormant, ε, κάποιοι από τους οποίους ήταν αδρανείς κτλ. Είχαμε συμφωνήσει με το ΕΛΚ να μην ψηφιστεί. Ε, τότε ας ψηφίσουμε να απορριφθεί λοιπόν. Αντί να αποσύρουμε τμήμα της συμβαστικής, ας το ψηφίσουμε, λοιπόν στο 3 υπέρ. Κατά, απεριφθεί, σαφές το αποτέλεσμα. Και νομίζω αυτή είναι η μόνη αλλαγή που είχα από τον κατάλογο. Προχωρώ γρήγορα κάποιες σελίδες, χάρη στις πολύ, στην πολύ καλή δουλειά των εισηγητών και σκιωδών. Και πάω στην 121 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, απεριφθεί. 143-144 υπέρ, κατά, απερίφθη, 149 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 150-153 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Απεριφθεί. Συμβαστική 9 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 179 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, ομού ψηφίζουμε την 190-198 υπέρ. Επαληθεύουμε παρακαλώ. 190 και 198 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται 22 της νομικής υπέρ κατά εγκρίνεται 200-201 υπέρ κατά εγκρίνεται απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά απορρίπτεται 13 της νομικής υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 204 με 207 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 221 με 224. Μόνο μία έχει αποσυρθεί, νομίζω. Πρέπει να ψηφίσουμε τι άλλε. Λοιπόν, οι διαγραφέ τη παραγράφου 9. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτονται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 233. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 19 της νομικής υπέρ. Κατά. να το επαληθεύσουμε όμως. 19 νομικής άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται 20 υπέρ 16 κατά. 236 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά. Απερίφθη. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο πάω λίγο πίσω. Την 236 την έχουμε εγκρίνει από ό,τι φαίνεται. Αφού εγκρίθηκε λοιπόν η συμβαστική 15 καταπίπτει. Από ό,τι λένε τα χαρτιά μου. Α, ηλεκτρονική ήταν η επιλήθευση. Ε. Ευχαριστώ να την ξανακάνουμε αν θέλετε. Με συγχωρείτε, είχαμε κάποιο λάθος, λέει η κυρία Πιετικάρεν, στον κατάλογο των ψηφοριών μας για τη 236. Δεν είμαστε υπέρ της ε, διαγραφής. Είμαστε κατά τη διαγραφή, για τον κατάλογο. Για τον κατάλογο. Ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν τάσσεται κατά της διαγραφής, κατά της τροπολογίας 236. ο πρόεδρος. Ε, φαντάζομαι ότι είναι ειλικρινέ το λάθο με την έννοια ότι δεν κάθεται κανεί να κάνει τόση δουλειά για τι συμβαστικέ ε, χωρί να θέλει να τι ψηφίσει. Επομένω. Λοιπόν, σα παρακαλώ, συνοηθείτε τουλάχιστον. Συμφωνήστε μεταξύ σα. Και σα παρακαλώ, σταματήστε να φωνάζετε. Κύριε Γκέπχαρτ, θέλω απλώ να επισημάνω ότι συνήθω δεν δέχομαι τέτοιε καταστάσει, αλλά αφού βλέπω ότι δεν είχε σημειώσει η γραμματεία το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του 236, δέχομαι να γίνει η επαλήθευση της ψηφοφορίας τώρα. Καλό είναι να συμφωνούν και οι σκιώδεις ηγητές. Η υπεύθυνη στάση αυτά υπαγορεύει. Ξανά κάνουμε λοιπόν την, την ψηφοφορία για το 236 θα είμαστε απόλυτος βέβαιοι έτσι για το τι ψηφίζουμε πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Και ψηφίζουμε την συμβαστική 15, να είμαστε βέβαιοι ότι την εγκρίνουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάω στη 253. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων Μετροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 255 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 του πολιτισμού καταπίπτει 256 υπέρ θα αρχίσει ψηφοφορία 256 παρακαλώ να επαληθεύσουμε πέρας απερίφθη με τρεις ψήφους τη φορά 6 τη Νομικής Επιτροπής υπέρ κατά εγκρίνεται 257 υπέρ κατά απερίφθη συμβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 273 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 του πολιτισμού υπέρ κατά εγκρίνεται 8 του πολιτισμού υπέρ κατά απερίφθη. 9 του πολιτισμού υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά απερίφθη. Καταπίπτουν οι επόμενες τμήμα της ε, συμβαστικής και τώρα πάμε 304 υπέρ όχι, καταπίπτει. Εφόσον εγκρίθηκε 290. Όχι απερίφθη, λέει ο πρόεδρος. 290. No, 290 was rejected. But 290 was rejected. Yeah. So, so, then we can. Yeah. So 304. Yeah. 304. 304. Κύριος Ταραμπέλα. Θα γλεντήσει υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Καλά να επαληθεύσουμε. 304 επαλήθευση. Άλλαξε γνώμη το έλκα από ό,τι φαίνεται. Πέρασε φορές εγκρίνεται. 305 και 13 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά εγκρίνεται 309-310 υπέρ Ας αρχίσει η ψηφοφορία. Απόρριπτε τρεις ψήφοι διαφορά. 19, συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 322 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 324 υπέρ. 324 υπέρ. Ας το επαληθεύσουμε, είναι λίγο ασαφές, αλλά μάλλον εγκρίνεται ίσα ίσα. 324 324 σας παρακαλώ ψηφίστε, ψηφίστε λίγο πιο γρήγορα. Πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 14 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 336 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 346 υπέρ. Κατά Απερίφθη. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 356 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 363-364 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά εγκρίνεται, τριά του πολιτισμού υπέρ, κατά εγκρίνεται, τέσσερα του πολιτισμού υπέρ, κατά εγκρίνεται, 23 της νομικών υπέρ, 23 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 17 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ, κατά εγκρίνεται, 18 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ, υπέρ, κατά... Δεν σε φες παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Και να σηκώνετε και τα χέρια το υπέρ, το και το κατά. Όχι εντάξει, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 24 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 367-368 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστικές 25 και 26 υπέρ. Κατά. εγκρίνονται. 34 της Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 375 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 385 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά εγκρίνεται 27 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά εγκρίνεται 17 της Επιτροπής Νομικών υπέρ. Κατά απερίφθη Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 406. Υπέρ. 406 υπέρ. Κατά. Κύριος Φόξ. Πρόεδρε, στην 406 λέει ότι αν εγκριθεί 410 καταπίπτει. Η 410 ήταν κομμάτι της συμβαστικής 28 που ψηφίσαμε. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος, άρα έχετε δίκιο. 406 την επαληθεύω όμως πάλι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, πολιτισμού 30, υπέρ κατά εγκρίνεται και 33 του πολιτισμού υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 18 ε, υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίθηκε, αλλά καλύτερα στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ 14 κατά. Συμβαστική τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ? Με την προφορική τροπολογία. Συμβαστική 30 με την προφορική. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Περνάμε στην... Στην τροπολογία 413. 413. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 400. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 415 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31 ε, ως προσθήκη της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 της Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 421. Καταπίπτει. 422. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 422. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά 18 προς 17. Τροπολογία 23 της Επιτροπής Πολιτισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων 25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 425. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 285 και 362. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 366. Ποιος είναι υπέρ. 366. Α, είναι πανομοιότυπη με τις προηγούμενες. Περνάμε στα θεωρώντας. 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Προς 18, μέχρι 18 πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 3 αποσύρεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, 12, 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 7 και 13. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογίες 15 και 16 υπέρ, κατά εγκρίνονται. Και περνάμε στα εκτιμώντας 19, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 86, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 45, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 46, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Α, ή μη, έχει αποσύρθει. Την αποσύρατε κυρία Πετικάνε. Α, η 48 έχει αποσυρθεί από την κυρία Πετικάνε. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 72, υπέρ. Τροπολογία 72, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 78, υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 78, άρχεται ψηφοφορία, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ και 14 κατά. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 80 παρακαλώ. Νομίζω ότι εγκρίνεται παρόλα αυτά. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλία. Άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 82. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 6α. Υπέρ. Κα... Υπέρ της 6α συμβαστικής τροπολογίας παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο της πρότασης. Ψηφίστε παρακαλώ όλοι. 34 χρειαζόμαστε και βλέπω 36 κάρτες έχουν μπει στο μηχάνημα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 32 ψήφισαν υπέρ, 3 κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Άσλι Φόξ. Και φυσικά ευχαριστούμε θερμά και τους σκιώδεις ηγητές. Θέλει κανείς το λόγο μήπως. Όχι. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα. Τη γνωμοδότηση που θα δώσουμε στις Επιτροπές Νομικών Υποθέσεων και Γυναικών με θέμα την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέση με εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Yeah. Απουσιάζει η συγγετρία κυρία Παραβάνοβα. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. μάντερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51 μάντερ υπερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 52-54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 55 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 και 56 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 6 και 56. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Διαδικαστικό. Η κυρία Χέντ. Μια στιγμή κύριε Πρόεδρε παρακαλώ. Περιμένετε λίγο. να ηρεμήσουμε λίγο και να κάνουμε λίγο ησυχία για να ακούμε τι ψηφίζουμε. Μα αυτό θα έκανα και εγώ, να ζητώ από όσους φεύγουν να, να μην μιλάνε ταυτόχρονα φεύγοντας, να αποχωρήσουν σιωπηρά. Αλλά αυτό δείχνει το, το ζωηρό ενδιαφέρον που προκάλεσε η προηγούμενη έκθεση του κ. Φόξ. Τροπολογία 7, Παρβάνοβα, τη ηγήτρια δηλαδή. Ποιο είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Παρακαλώ ψηφίστε λίγο πιο γρήγορα. Εγκρίνεται 22 προς 10. Τροπολογία 57 του κ. Μάντερς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58 της κυρίας Χέντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 της κυρίας Χέντ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 και 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 63. Ποιος είναι υπέρ. Συγγνώμη, 61 λέει ο πρόεδρος. Πήδηξα μία. 61. Ποιος είναι υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 61. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για έλεγχο, γιατί βλέπω πολύ το σχετισμό δυνάμενο. Παρακαλώ ψηφίστε γρήγορα για την 62. Τέλος ψηφοφορίας. 32 ψηφίζουν, 20 προς 10 εγκρίνεται. Η 63 καταπίπτει. 64 της κυρίας Χέντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 65 του κυρίου Μάντερς υπέρ κατά. Και αυτή απορρίπτεται. 66 της κυρίας Χέντ υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 66. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Παίρνουμε στα 10 τροπολογία υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 με ψηφοφορία κατά τμήματα. Βλέπετε το πρώτο τμήμα, χωρίς το περιλαμβάνοντας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέσσερις ψηφίζουν εδώ. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Γιατί 13 κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 13 παρακαλώ. Ή μάλλον εγκρίνεται. Για να δούμε. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή με την ίδια διαφορά. Τροπολογία 2 της εισηγητρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 με ψηφοφορία κατά τμήματα, το ίδιο πάλι. Το πρώτο τμήμα χωρίς το όπως η ΕΚΤ, ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται με διαφορά και το δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται με, τις ίδιες, με την ίδια διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4 της κυρίας Παρβάνοβα της ηγετρίας. 31 μόνο ψηφίζουν οι 33. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. 15 προς 18. Τροπολογία 22 της κυρίας Λεγκρίπ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Παρβάνοβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Μάντερς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 26. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 17 προς 15. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 28 με προφορική τροπολογία, τη διαβάζετε δίπλα, της κυρίας Χέντ, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 29 με προφορική τροπολογία, υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29, μάλλον απορρίπτεται όμως. Τέλος ψηφοφορίας. όχι. Εγκρίνεται τελικά με μία ψήφο διαφορά. 17 υπέρ, 16 κατά. Συμβαστική τροπολογία 4. Α, συγγνώμη, 30 πρώτα τροπολογία της κυρίας Head. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οι φιλελεύθεροι ψηφίζουν. Δεν το γνωρίζουμε. Παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί νομίζω ότι οι φιλελεύθεροι δεν ψήφισαν. Τροπολογία 30 ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. 32 ψηφίζουν μόνο, 18 υπέρ, 14 κατά. Τελικά αποφάσισαν να υπερψηφίσουν οι φιλελεύθεροι. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34 το κύριο Μάντερς, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά απορρίπτεται 39 υπέρ κατά απορρίπτεται 40 υπέρ κατά απορρίπτεται 41 υπέρ κατά απορρίπτεται 42 υπέρ κατά απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος ηλεκτρονικός έλεγχος για την 42 32 ψηφίζουν μόνο. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται, εγκρίνεται. Ευχαριστώ που μου το επισημάνατε. 18 υπέρ, 14 κατά. 43 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται και 44 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 27 υπέρ 3 κατά 3 αποχές. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Παραβάνοβα. Έχουμε τώρα δύο σύντομες ψηφοφορίες. Παρακαλώ ε, μείνετε στην αίθουσα γιατί θέλουμε κάποιες πλειοψηφίες να συγκεντρώσουμε. Έχουμε το διορθωτικό δεύτερης ανάγνωσης της πρότασης Κρόιτσμαν για την τελωνική εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα πρακτικά, το κείμενο της συνδιαλλαγής Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ, μία ψήφος κατά, εγκρίνεται το κείμενο. Και ένα διορθωτικό στην οδηγία για τα παιχνίδια, για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Διανατάσεις χειρός ή θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το διορθωτικό για την έκθεση για την ασφάλεια των παιχνιδιών χρειάστηκε το διορθωτικό μετά από συζήτηση με τους ηγετές, άρχεται η ψηφοφορία για το διορθωτικό της ε, έκθεσης για τα παιχνίδια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τεχνική αλλαγή στην οδηγία για τα παιχνίδια. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 30 υπέρ ψηφί Σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και μπορούμε να περάσουμε και νωρίτερα από το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα στην έκθεση για το δίκαιο των πωλήσεων. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, πεντάλεπτο, ώστε όσοι θέλουν να φύγουν να αποχωρήσουν και να περάσουμε μετά στο κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Άλλωστε παραβρίσκονται και οι δύο εισηγητέ. Και ο κύριο Φόκ. Thank Ξαναρχίζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να προχωρήσουμε γρήγορα. Μια και τελειώσαμε πιο νωρί τι ε, ψηφοφορίε, θα μπορούσα να σα δώσω ακόμη ένα τέταρτο, αλλά α ξεκινήσουμε το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Έχουμε δύο εισηγητέ, ε, η κυρία Γκέπχαρτ και άλλος ένας που δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Ο Κρόιτσμαν, η κυρία Ρούλε, ο Άσλι Φόξ ήταν οι σκιώδεις εισηγητές. Δεν βλέπω τους υπόλοιπους. Ο κύριος Μάιερ ε, από την Επιτροπή είναι εδώ. Είναι τακτικός επισκέπτης στην Επιτροπή μας. Είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπρόσωπο. Ε, σίγουρα θα του δώσουμε και λίγο χρόνο για να απαντήσει στις τροπολογίε. Δεν ξέρω ποιο θέλει να πάρει πρώτο το λόγο. Ποιο από του δύο εισηγητέ. Ο κύριος Μάιερ ή η κυρία Γκέπχαρτ. Α, η κυρία Γκέπχαρτ είναι τόσο πολύ ευγενική, προσφέρει το, την πρωτοκαθεδρία στον κύριο Μάιερ. Πρώτα ο κύριος Μάιερ λοιπόν, μετά η κυρία Γκέπχαρτ, μετά οι υπόλοιποι ισχυώδεις εισηγητές και οποιοδήποτε άλλο θέλει να συνεισφέρει εν συνεχεία. Και ευχαριστώ κύριε ε, Γκέπχαρτ που μου δίνετε το χρόνο σας. Μετά στις απαντήσεις θα αλλάξουμε σειρά. Έχουμε λοιπόν ε, τις ε, τροπολογίες, συζήτηση για τις τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ε, επί της αρχής έχουμε ήδη ασχοληθεί με το θέμα και μάλιστα σε διάφορες επιτροπές. Έχει ήδη ψηφίσει επί της ουσίας επί του βασικού ερωτήματος η Ολομέλεια, δηλαδή ποια θα πρέπει να είναι η μορφή ε, του δικαίου των πωλήσεων που θα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με μεγάλη, με βήτατη πλειοψηφία επέλεξε το ενδοτικό ή δυνητικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι τις έχουν διατυπώσει. Και πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές που προτιμούν οι δύο ε, αλλά οι οποίες είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Δηλαδή καταρχήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε συμβασμούς σε ε, ορισμένα μεμονωμένα αισθήματα ναι, αλλά όχι επί της αρχής. Θα σας εξηγήσω όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Η Εύελιν και κάποιοι άλλοι θα ήθελαν αντί για το ενδοτικό σύστημα να ζητήσουν την διεύρυνση του αρχικού ε, νομοθετήματος της οδηγίας για το καταναλωτικό δίκαιο και μια διεύρυνση άλλο συνάδελφος της οδηγίας του 99 για τα καταναλωτικά αγαθά με τις εγγυήσει και την ε, διάρκεια ζωής των προϊόντων με παραπομπή για την, στην οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου και προσδιορισμό των προϋποθέσεων για τα προϊόντα τα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, στην ε, σχετική οδηγία του 2009. Μια έκθεση της μελέτη μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτείται ως εκ τούτου για τον κύκλο ζωής των προϊόντων και εγώ θεωρώ ότι μπορούμε αυτή τη βάση, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κοινό εμπορικό δίκαιο, να την αξιοποιήσουμε αντί για ένα ενδοτικό σύστημα ή δυνητικό εργαλείο, ε, για να τροποποιήσουμε τις υφιστάμενες οδηγίες, λένε κάποιοι. Εγώ όμως νομίζω ότι νομικά δεν υπάρχει δυνατότητα, δεδομένου ότι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι εμείς δεν είμαστε εκτελεστική εξουσία. Αυτά τα έχει και είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί λοιπόν μόνο με έκθεση πρωτοβουλία θα μπορούσαμε να τυπώσουμε αυτέ μα τι θέσει και προτιμήσει, αλλά όχι με τη μορφή μια συγκεκριμένη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για μένα το κύριο ε, ζήτημα είναι αν θέλουμε ένα δυνητικό σύστημα ή ένα υποχρεωτικό. Εγώ προτιμώ το δυνητικό, η Εύελιν δεν το θέλει, άρα ω εκ τούτου για να είναι συνεπή με τι θέσει θα πρέπει να απορρίψει τι προτάσει τη Επιτροπή. Αλλά πάντω δεν μπορούμε να ζητήσουμε ή να απαιτήσουμε τελείω διαφορετικά πράγματα ή την προσθήκη ε, άρθρων, όπω θα λέγαμε στην Γερμανία, δηλαδή τι τροπολογίε αυτέ, οι οποίε θα άλλαζαν ουσιαστικά το κείμενο. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν του συναδέλφου που έχουν καταθέσει τροπολογίε, τι γνώμη έχουν σε αυτά. Ω προ το περιεχόμενο των τροπολογιών. Πέραν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο των πολλών συναδέλφων, ανδρών και γυναικών που έχουν κάνει αποκοδομητικέ προτάσεις, βλέπω ενδιαφέρουσες προτάσεις και για το όσο έχουν πει κύριοι Όπερ Μάιερ, Φραντσμαν, Ρέπο, ε, προ, ε, προτάσεις δηλαδή οι οποίες μπορούν να εγγραφούν μέσα στο σύστημα. Και βεβαίω μπορούμε να διατυπώσουμε συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά για αυτέ τι τροπολογίε βλέπω ότι είναι δυνατόν να ενσωματωθούν με κάποιον τρόπο. Το θέμα όμω τη ολικά διαφορετική προσέγγιση στο θέμα αυτό, πώ θα το επιλύσουμε. Αυτό νομίζω θα χρειαστεί να το συστήσουμε σε μια ειδική συνεδρίαση οι δύο συνεισηγητέ. Είπα ήδη και θα πρέπει να το ε, υπογραμμίσω μια φορά ακόμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επί της αρχής υποστηρίξει την ιδέα του, της ε, δυνητικής εισπαγωγής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό το απορρίπτει η Γερμανική κάτω βουλή, ενώ το Bundesrat βλέπουμε να επιβληθεί θέλει να επιβληθεί το δυνατικό δίκαιο, όπως ε, άλλωστε και η Εύελιν Γκέρπχαρτ, δεδομένου ότι οι εκπρόσωποι της δικής της πολιτικής ομάδας και πολιτικού κόμματος επικρατούν εκεί τώρα. Τέλος πάντων σε αυτό επιμένετε, τι να πω εγώ. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας, τα δύο, ε, ε οι δύο ασυμφιλίωτες διαφορές, ε, αγεφύρωτες διαφορές που θα πρέπει όμως κάπως να ε, λύσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Κάπως πρέπει να τα συμφιλιώσουμε. Αλλά πολύ σωστά παρουσιάσατε ξεκάθαρα τις διαφορές αυτές. Ε, μας είπατε ποια είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Στη χώρα μου έχουμε καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ για να μην δώσω περιθώριο σε εσφαλμένες εντυπώσεις. Όταν ε, τοποθετήθηκε το γερμανικό Bundesrat, εμεί δεν είχαμε ακόμα μέσα την ε, πλειοψηφία οι σοσιαλδημοκράτες ε, στου κόλπου του. Μην δοθεί εντύπωση δηλαδή ότι μόνο οι σοσιαλδημοκράτες επιδιώκουν αυτή τη λύση του δυνητικού δικαίου. Όλες οι ομάδες στη Γερμανία είχαν συμφωνήσει κατά του δυνητικού συστήματος και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένα σαφέστατο μήνυμα και θα έπρεπε να είναι ένα σαφέστατο μήνυμα προς τη γερμανική κυβέρνηση. Και κάτι ακόμη. Η έκθεση Wallis, για την οποία λέγεται πάντοτε ότι ε, έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώσει μέσω της εκθέσεως αυτής ότι προτιμάει το δυνητικό σύστημα. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την εκθέση βόλης. Διότι μπορεί να λέγεται εκεί ότι ε, θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο σύστημα και θα έπρεπε να συζητηθεί, αλλά από την άλλη καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση επιπτώσεων και να εξετάσει με μεγάλη ακρίβεια τι είδου επιπτώσει μπορεί να φέρει αυτό το σύστημα και ταυτόχρονα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει τα λοιπά υφιστάμενα συστήματα. Οι δε υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέτασαν αυτή η μελέτη επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαν ε, ότι μεθοδολογικά έχει ε, ακολουθήσει τη σωστή μεθοδολογία, αλλά παραμένουν στα αποτελέσματα κάποια σημαντικά προβλήματα και ως εκ τούτου τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει αυτή η μέρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι θεμελιωμένα, δεν ε, εδράζονται σε γερά θεμέλια και ως εκ τούτου αμφισβητούνται. Και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ίδιες ε, είπαν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ε, σε επίπεδο αυτής της μελέτης ε, επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ότι ξεκίνησε με προσέγγιση το δυνητικό ε, σύστημα χωρίς να επεξεργαστεί επαρκώς τα υπόλοιπα προσφερόμενα συστήματα, ώστε να δει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός. Και εν προκειμένου δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν κάνουμε νομοθετήματα, όταν συντάσσουμε, καταρτίζουμε νόμους, θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας απόλυτα απτά και θεμελιωμένα επιχειρήματα, μια γερή βάση δηλαδή, πάνω στην οποία να μπορούμε να στηριχθούμε για τις τροπολογίες. Βλέπω μια σειρά από καλές τροπολογίες και τι θα τα πω, είπε ο Χανς Πέτερ. Εγώ τις δέχομαι, τις εξετάζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα όλες τις τροπολογίες, ούτε ξεφεύγω σε τέτοιου είδους υφολογικές ε, διαφοροποιήσεις ως προς τη σοβαρότητα των τροπολογιών, ώστε να προσπαθώ να γελιοποιήσω κάποιες χάρτες Πέτερ. Τις παίρνω όλες πολύ στα σοβαρά και τις εξετάζω όλες με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ο Γομπέχος Φόχ στις ε, τροπολογίες του ε, αναφέρεται σε κάτι που βρίσκω πολύ σημαντικό, την αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεν μπορούμε να τα λησμονήσουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε και νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα σημείο ε, εκκίνησης που θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε. Και επίσης για, κυρία, για τον κύριο Ρέπο ε, είπατε κύριε Χάνς Πέτερ Μάιερ ότι θα κάνετε εσείς ε, δεκτές τροπολογίες που αφορούν το δυνητικό σύστημα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία εμείς μπορούμε να δεχθούμε, αλλά μην σκέφτεσαι ότι ο Νίκτρο Ρέπο ή ο Γιωβάιναν είναι υπέρ του δυνητικού συστήματος, γιατί μου το έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν το υποστηρίζουν. Απλώς θέλουν ε, να εισαγάγουν κάποια στοιχεία τα οποία εγώ προσωπικώς δεν έχω ε, προβλέψει. Κατά τα άλλα συμφωνούν με τις δικές μου τροπολογίες, απλώς δεν τις επαναλαμβάνουν και αυτό το λέω για να καταστεί σαφές και να μην ακούγονται παραμυθάκια και μύθοι δεξιά-αριστερά για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα από σένα, Χανισπέτσα. Μία σειρά από τροπολογίες τις οποίες απλά και μόνο δεν μπορώ να υποστηρίξω, είναι η Μάιερ Κρόιτσμαν, Κόλιν Μάλεν, που βεβαίως ε, θέλουν το δυνητικό σύστημα και δεν δέχονται που δεν είναι, δεν δέχομαι που δεν είναι τις τροπολογίες Κρότσμαν που επιδιώκουν, ε, που οδηγούν στην ε, υποβάθμιση της προστασίας του καταναλωτή και ξεπερνούν αυτό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά υποβαθμίζουν το πραγματικό, το ουσιαστικό ε, δίκαιο προστασία του καταναλωτή, όπω αυτό ισχύει και στα κράτη-μέλη. Και ιδιαίτερα την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, αυτή που είχαμε εγκρίνει το 2011. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε πουθενή. Ούτε έχω ούτε η ομάδα μου. Κύριε Κρόιτσμαν, θα σας πω ξεκάθαρα όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερη προστασία του καταναλωτή, δεν μπορούμε να ε, απεισχνάσουμε τόσο πολύ την προστασία του καταναλωτή που υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι παράδεκτο αυτό για μένα. Επίσης, για τις τροπολογίες Fox, στο βαθμό που δεν τις έχουμε συντάξει από κοινού και τις υπόλοιπες μπορώ να τις δεχθώ, απλώς θα ήθελα με θετικό πνεύμα λίγο να ξανασκεφτώ μια ιδέα από αυτές. Γιατί για μένα η πρόταση είχε σαν στόχο την ελάχιστη ε, εναρμόνιση και γι' αυτό κύριε Στορμένη θα ήθελα να παρακαλέσω να μην μιλάτε μόνο για σε ελάχιστους όρους, όπως προσπαθείτε εσείς να ε, περιγράψετε, ελάχιστη εναρμόνιση σημαίνει ελάχιστος κοινό παρονομαστής, όχι οι λιγότεροι δυνατοί κανόνες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότεροι, ώστε να έχουμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Ο κύριος Ροσφόρ προσπαθεί να διατυπώσει με τις τροπολογίες του στο δυνατόν, ε, τη διεκδίκηση για μια στο δυνατόν μέγιστη τροπολογία, αυτή την ε, εναρμόνιση, αυτή την τροπολογία λοιπόν εγώ μπορώ να τη δεχθώ στο βαθμό που σε ορισμένους τομείς μπορεί όντως να εξασφαλίσει πιο προοδευτικό δίκαιο, κοινό δίκαιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό νομίζω ότι θα ήταν κάτι το θετικό, γιατί εν τέλει θα σήμαινε ότι έχουμε ακολουθήσει έναν δρόμο, όπως και με την οδηγία για, τον, ε, για το δικαίωμα του καταναλωτή που συντάξαμε στον κύριο Σφάπ, μια οδηγία ε, μεικτή που θα επιλέγει το δρόμο της ε, μεγίστης εναρμόνισης εκεί όπου αυτή είναι δυνατή και η δάλος όπου δεν είναι δυνατή της ελάχιστης εναρμόνισης σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος. Και πριν τελειώσω θα ήθελα να παρακαλέσω μια και είδα ότι είναι παρόν και το Συμβούλιο και προσωπείται σήμερα εδώ και μια και ο κύριος ε, λένε ε, εχθέ μου επέτρεψε να παρουσιάσω τι τροπολογίε μου για την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, όπου μου είπε ο κύριο Λένε ότι το Συμβούλιο έχει επιλέξει εν τέλει το δυνητικό σύστημα, απερίφραστα, και ότι η Λιθουανική Προεδρία σκοπεύει να ε, καταστήσει το ζήτημα αυτό με την επιλογή του δυνητικού συστήματος ε, προτεραιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την Ιρλανδική Προεδρία να μας πει ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Μάλκομ θα θυμάσαι κι εσύ φαντάζομαι ότι είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό των Οικονομικών τη Λιθουανίας ο οποίο μα είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν προτεραιότητα τη Προεδρία του και ότι δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να, να προωθήσει αυτό το φάκελο. Τώρα βλέπω να ακούγονται διαφορετικέ δηλώσει. Μια και έχουμε εδώ λοιπόν την Ιρλανδική Προεδρία, α μα πούνε, α μα διαφωτίσουν, α μα πούνε ποια είναι η κατάσταση ακριβώ. Και πριν να σταματήσω θα επισημάνω και το εξής. Ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αισθάνομαι μεγάλη δυσφορία ως προς την στάση και τη μεθοδολογία που έχουν επιλέξει η Επιτροπή των Νομικών, ο Χάνς Πέτερ Μάιερ και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή βλέπω μία διάκριση μεταξύ του υπερσυνοριακού και του μη υπερσυνοριακού εμπορίου και βλέπω και διάκριση μεταξύ κατηγοριών προϊόντων. Και μετά βλέπω και στο άρθρο 13 ότι προβλέπεται η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη, εφόσον το επιθυμούν, και στους τομείς στους οποίους δεν υπάρχει δυνητικό σύστημα σε ευρωπαϊκό δίκαιο, να εισαγάγουν το δυνητικό αυτό δίκαιο στην εσωτερική τους αγορά, για τις εσωτερικές τους συναλλαγές. Αυτό πολύ φοβούμαι ότι θα μας οδηγήσει στο απόλυτο χάος ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να ξεχωρίσουν τι ισχύει, τι δεν ισχύει, δεν μπορούν να βρουν την άκρη. Γιατί ένας ε, εκπρόσωπος του direct marketing από τη Γαλλία που συνάντησε την Δευτέρα μου εξήγησε ότι είναι πολύ δύσκολο το πρότυπο αυτό το δυνητικό και μου είπε ότι επαληθεύσαν ε, πώς μπορεί ο νέος καταναλωτής, ο νεαρός καταναλωτής να μπει μέσα στην αγορά και αυτό που παρατηρείται ως φαινόμενο είναι ότι ο νέος καταναλωτής πηγαίνει στο κατάστημα, βλέπει το προϊόν του, αλλά δεν το αγοράζει εκεί, το αγοράζει μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο, ότι είναι όλο και πιο δικτυωμένος ο νέος καταναλωτής, βρίσκεται μέσα στο μαγαζί, βλέπει το προϊόν και με, με το άλλο χέρι ε, παίρνει το κινητό του και κάνει την παραγγελία μέσω του διαδικτύου. Και λέει, και πρέπει να είναι σε θέση να πει ότι να τώρα βρίσκομαι στο μαγαζί και άρα αγοράζω με βάση το γερμανικό ή το γαλλικό δίκαιο ότι ισχύει, αλλά μέσω του διαδικτύου και μέσω του κινητού μου μπορώ να έχω ένα φθηνότερο προϊόν με ένα δυνητικό σύστημα ευρωπαϊκού δικαίου, για το οποίο όμω δεν γνωρίζω τελικά τι ισχύει και τι αποτέλεσμα θα βγει και ποια θα είναι εφαρμοσόμενη διάταξη. Ε, φανταστείτε τώρα του νέου καταναλωτέ τη Ευρώπη, του νεαρού καταναλωτέ τη Ευρώπη, που είναι συνδεδεμένοι με όλα τα ε, μέσα μαζική επικοινωνία και που μπορούν να αξιοποιούν κάθε δυνατότητα τη δικτύωση, να βρίσκονται μέσα σε αυτό το δίλημα. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε αυτό το δυνητικό σύστημα μπορεί να έχει βέβαια κάποιο πλεονέκτημα. Δημιουργία θέσεων εργασία για δικηγόρου. Αλλά μόνο αυτό. Τίποτε άλλο και καμία σχέση με ασφάλεια δικαίου που επιδιώκουμε. Θα επανέλθουμε σε αυτό όταν ξαναδώσω τους, τους συζητητές το λόγο για να το σχολιάσουν. Κύριε Σάνς Πέτερ αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και το, το, το ξέρω και εγώ έχω δει ότι πηγαίνει κανείς σε ένα μαγαζί και κοιτάει ταυτόχρονα τις τιμές στο ίντερνετ γιατί εκεί μπορεί να είναι πιο φτηνά τα προϊόντα, δεν υπάρχουν έξοδα αποθήκευσης και το καθεξής. Αλλά μετά έρχεται μια προσφορά από τη Λιθουανία ή την Αγγλία ή τη Βρετανία ή τη Γαλλία. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Διότι η επιλογή αυτή που θα έχει μέσα στο διαδίκτυο υπάγεται σε τρία διαφορετικά δίκαια και αυτά θα πρέπει να ε, δει αν θα εφαρμοστούν και όχι το γερμανικό ή το ισπανικό ανάλογα που θα βρίσκεται. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε, λέει η κυρία Γκέπχαρτ, ότι υπάρχει ο κανονισμός Ρώμη 1 όπου τα δικαιώματα του καταναλωτή είναι αυτά τα οποία ε, εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα και έχουν την προτεραιότητα, πράγμα το οποίο θα αναιρέσει το δυνητικό σύστημα. Αυτά είναι ζητήματα που θέλαμε να συζητήσαμε όταν κάναμε την ε, προηγούμενη συζήτηση για τις αρχές. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και τη μελέτη αντικτύπου. Πρέπει τώρα όμως να ακούσω τους υπόλοιπους ε, σκιώδης συζητητές, ο κύριος Κρόιτσμαν και ο κύριος Φόξ μετά. Ναι, να δούμε όμως και τι θέλουμε κυρία Γκέπχαρτ. Αυτό που, έχουμε επιτύχει, αυτό που έχουμε επιτύχει και εκεί που έχουμε φτάσει στην εσωτερική αγορά ή θέλουμε να πάμε και λίγο παραπέρα. Και θα σας ε, επαναφέρω στο θέμα των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Με πρώτη παρατήρηση ότι ακούσαμε, το είπε και ο κύριος Μάιερ, ποια είναι τα επιχειρήματα, τα έχουμε δει και στην πράξη όταν ο κύριος Σφάπη θέλησε να ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες και στάσεις και κουλτούρες. Στο θέμα το δυνητικό λοιπόν μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο, γενικό εμπορικό δίκαιο με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτό μπορεί να μα το επιτρέψει το δυνητικό σύστημα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι υποχρεωμένη καμιά επιχείρηση να το ακολουθήσει. Άρα, βγάζουμε τον παράγοντα κίνδυνο λέγοντας φτιάχνουμε μια μεγάλη αγορά και η προστασία του καταναλωτή, η ενισχυμένη προστασία του καταναλωτή είναι προς το συμφέρον της μεγάλης αγοράς. Εκεί θα πρέπει να σταθμίσω εάν θέλω να προστατέψω και την επιχείρηση ή να την έκθεσω σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Για να δούμε λοιπόν στη Γαλλία ή τη Γερμανία. Μια μεγάλη αγορά. η οποία μπορεί να μην ενδιαφέρει καθόλου, να μην ενδιαφέρεται καθόλου να πουλήσει στο Λουξεμβούργο τη Λετωνία την ε, Εσθονία γιατί είναι μικρές αγορές. Άρα όταν έρθει η ώρα για υψηλής, ε, υψηλών απαιτήσεων προδιαγραφές για το καταναλωτή, απλώς δεν θα πουλήσει στις αγορές αυτές γιατί δεν θα τον ενδιαφέρει. Πρέπει λοιπόν τον καταναλωτή να τον δούμε σαν ένα όλο, ο οποίος θα μπορεί και να επιλέξει εάν θέλει να αγοράσει ή όχι και αν θέλει την υψηλότερη προστασία των δικαιωμάτων του. Ε, νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να, μπορούμε να ακολουθήσουμε το δυνητικό σύστημα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι δεν αμφισβητούνται τα δικαιώματα του καταναλωτή στην υπόθεση αυτή. Βεβαίως έχετε δίκαιο ότι δεν μπορούμε να ε, οπισθοδρομήσουμε ως προς τη Γενική Οδηγία περί δικαιωμάτων του καταναλωτού. Σε αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ε, επιδείνωση των συνθήκων. Αλλά εκεί όπου υπάρχει μία πρόθεση για ενίσχυση των δικαιωμάτων της προστασίας του καταναλωτή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λογικής εφαρμογής, είτε πρόκειται για δυνητικό είτε για μη δυνητικό σύστημα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα συμφέρον ο καταναλωτής να τον προστατεύουμε με μία νομοθεσία την οποία απλώς και μόνο δεν θα εφαρμόσει η επιχείρηση, δεν θα την αξιοποιήσει λύση. Γιατί τότε έχουμε ουσιαστικά προστατέψει τον καταναλωτή στο μεγαλύτερο κράτος μέλος που μπορεί να έχει την πρόσβαση αυτή, ενώ στο μικρότερο κράτος μέλος να την έχει, γιατί το είπε και ο κύριο Μάγερ ότι μπορεί να πάει στο μαγαζί και να δει το προϊόν στο κατάστημα, αλλά να προτιμήσει να αγοράσει από το διαδίκτυο γιατί είναι πιο φθηνό εκεί. Ε, αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσφέρουμε σε δυνατότητα όχι μόνο στο Γερμανό, αλλά σε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνω και εγώ στη Γερμανία. Μπορώ να πάω, όχι εγώ, τα παιδιά μου μάλλον, ε, μπορώ να πάω στο κατάστημα να κοιτάξω το προϊόν ε, ε, να το πιάσω στα χέρια μου και μετά να το αγοράσω από το ίντερνετ. Γιατί είναι λίγο φθηνότερο. Από την άλλη, πολλές φορές προτιμώ να πάω στο κατάστημα και να αγοράσω, και εσύ είναι λίγο φθηνότερο το διαδικτυακό κατάστημα, διότι μπορώ να έχω την επικοινωνία με τον ε, πολιτή, μπορώ να ρωτήσω τις πληροφορίες που χρειάζομαι, μπορώ να έχω καλύτερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση όπου δεν λειτουργεί όπως ή δεν μπορώ να το κάνω να λειτουργήσει, το μηχάνημα κτλ. Άρα λοιπόν ε, ένα προϊόν το οποίο δεν χρειάζεται τεχνική υποστήριξη μπορεί να απολυθεί πιο εύκολα στο ίντερνετ ε, γιατί είναι απευθείας ε, καταναλώσιμο, δεν χρειάζεται οδηγίες χρήσεως κτλ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αποκλείεται η αγορά και στο κατάστημα και το ότι δίνουμε ένα δυνητικό σύστημα δεν σημαίνει ότι επιδεινώνουμε τις συνθήκες προστασίας για τον καταναλωτή. Γνωρίζουμε πολύ καλά εξάλλου ποια είναι η τοποθέτηση και της γερμανικής, ε, του γερμανικού οικονομικού κλάδου, της γερμανικής βιομηχανίας που τάσετε κατά αυτής της υποχρεωτικής εισαγωγής όπως τη ζητάτε εσείς. Γιατί λένε ότι θα θέλει να αγοράσει κανείς. Μα ναι, αλλά ένα λεπτό, κύριε Γκέπχαρτ, αυτό ακριβώ θα είναι το πρόβλημα. Ότι θα θεσπιστεί μία νομοθεσία η οποία δεν θα φέρνει αποτέλεσμα, δεν θα εφαρμόζεται από κανέναν. Και αυτό δεν είναι προ το συμφέρον μα. Ξέρω ότι η πολιτική μου ομάδα στο Βερολίνο έχει επιφυλάξει προς το δυνητικό σύστημα, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε σε μια προσφορά, μια προσφορά που πρέπει να αξιοποιήσουμε και έτσι... Όπω είπατε, δεν επιδεινώνουμε τι συνθήκε σε σχέση με τα όσα προβλέπει η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε με την δυνατότητα προσφοράς μιας, ε, με τη δυνατότητα να υπάρχει μια προσφορά ικανοποιητική για τον καταναλωτή χωρίς βέβαια να επιδεινώνεται, να επιδεινώνεται το επίπεδο των δικαιωμάτων του. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω στον κύριο Κρόιτσμαν ότι εγώ θέλω να υπάρξει προδό στην ενιαία αγορά. Το ξέρετε ότι το θέλω. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό χάρη σε αυτή την πρόταση. Αντίθετα, είναι η παναχώρηση Μήπως είναι προσωπική φιλοδοξία της ε, Vivian Redding παρά προσπάθεια προστασίας των καταναλωτών. Είμαι αντίθετος, όπως ξέρετε, σε αυτή την πρόταση. Είμαι... Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ε, ωφέλη για τα κράτη-μέλη, τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις. Ε, οι εμπλεκόμενοι, ε, κυρία Γκέφχαρτ, εγώ, αντίθετα από εσά, πιστεύω ότι είναι αντίθετη σε αυτή την πρόταση. Γιατί σπαταλούμε χρόνο, ενώ θα έπρεπε να δούμε τους διαφορετικούς κανόνες ε, της ε, διαφήμισης, ε, σωστά ενδικά μέσα κτλ. Αυτά πρέπει να, αυτά πρέπει να προωθήσουμε. Γιατί με αυτή την πρόταση δημιουργείται ανασφάλεια ως προς την ερμηνεία του δικαίου, δημιουργεί επιπλέον κόστος και τελικά θα το φέρουν αυτό οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Και έχω μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση και την εξετάζουμε αυτή η πρόταση, ενώ στην παραδεχτήκατε ότι η δική σας μελέτη αντικτύπου ήταν προβληματική. Λοιπόν, αυτές είναι οι κάποιες αρχές, κάποια δεδομένα. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόταση ρεαλιστικά. Εγώ προσπάθησα να τη δω ρεαλιστικά μέσω των τροπολογιών μου. Παρότι θεωρώ ότι είναι ρηξικέλευτη προσέγγιση, ε, υποστηρίζω την κυρία Γκέπχαρτ που θέλει να αλλάξει η πρόταση αυτή και να γίνει οδηγία. Ανησυχώ λιγάκι για την έλλειψη πληροφοριών που έχουμε για τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της ε, αλλαγής και πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μία μελέτη αντικτύπου για τα ωφέλη ε, εφόσον γίνει αυτή η πρόταση οδηγία. Ε, φαντάζομαι θα το κάνει, γιατί νομίζω ότι έχει αποφασίσει ποια πορεία θα πάρει και ό,τι και στοιχεία και να τις δώσουμε θα επιμείνει ακάθεκτη. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να δούμε, ούτω ώστε να υπάρξει ισορροπία ξανά σε αυτή την πρόταση ε, υπέρ των καταναλωτών. Έχω, για το, έχω τροπολογίες για τα, τις μοντέρνες συμβάσεις, ε, τις τυποποιημένες ε, προϋποθέσεις και όρους. Η προσέγγιση στα ένδικα μέσα θα οδηγήσει σε φοβερή αλλαγή απαράδεκτη για το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. τώρα αν εμείς έχουμε πρόβλημα ε, στην αγορά, ε, βραχυπρόθεσμα μπορούμε να προσφύγουμε. Ενώ ε, αυτό το βραχυπρόθεσμο δικαίωμα προσφυγής θα χαθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα ε, ενδίκων μέσω εγχώριου και θα δημιουργηθεί ανασφάλεια για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που θα θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Γι, γι αυτό μαζί με την κυρία Γκέμπχαρτ, έχω υποβάλει τροπολογίες ε, για τα μοντέλα ε, συμβάσεων ως εναλλακτικό τρόπο, γιατί τα ένδικα μέσα που προτείνονται δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με την οδηγία ε, προστασία των καταναλωτών, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε κάποιο επίπεδο εναρμόνιση. Και οι καταναλωτέ και οι επιχειρήσει θα επωφεληθούν από αυτέ τι συμβάσει που θα βασίζονται στο κεκτημένο για του καταναλωτέ. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν αυτέ τι τροπολογίε που θέλουν να εξασφαλίσουν μια νομική εναρμόνιση ε, με σκοπό το υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Θα ισχύει για όλε τι αγορέ, ούτω ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά και παρόλα, παράλληλα θα υπάρχει ισοτιμία ε, για τι επιχειρήσει ε, σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, για το Σύμβουλο δεν υπάρχει συνένεση για αυτήν την πρόταση, ε, είναι αντίθετη και συμφωνώ και κάνω έκκληση και παρατρύνω τους Ιρλανδούς να μην προωθήσουν αυτήν την πρόταση. Σας ευχαριστώ όλους. Προ, ε, υποσχέθηκα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν χρόνο για να απαντήσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι και υπερβολικά γενναιόδωρος, γιατί έχουμε ακόμα και το θέμα του καπνού. Και σε αυτό το θέμα έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Αν η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να απαντήσει, φυσικά μπορεί να το κάνει. Αλλιώ θεωρώ ότι άκουσαν πολύ προσεκτικά τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Αλλά τώρα καλώ τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι άποψη έχει για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής και οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλει να θέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω δύο λόγια καταρχήν για ένα σημείο που ακούστηκε από πολλούς ε, ευρωβουλευτές για τη μελέτη αντικτύπου. Και συνεχεία να πω δύο λόγια για το θέμα της φύσης ε, του μέσου, την εναρμόνιση, τι είδου ε, σε εναρμόνιση προωθεί αυτό το μέσο, αυτό το κείμενο και να σχολιάσω το πρακτικό παράδειγμα της κυρίας Κέφχαρτ. Ήταν θαυμάσιο παράδειγμα για να σας δείξω μέσω ενός παραδείγματος πώς λειτουργεί η πρόταση στην πράξη. Πολύ σύντομα. Για τη μελέτη αντικτύπου καταρχάς. Καταρχάς. Και απαντώντας στον κύριο Φόξ. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε, δεν παραδεχόμαστε ότι η μελέτη που μα ήταν προβληματική. Αντίθετα, είμαστε περήφανοι και θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αυτή η μελέτη. Σε ό,τι αφορά τι επικρίσει τη κυρία Γκέπχαρτ. Είπε ότι δεν ε, υπάρχουν σχετικές, ε, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τα θεμέλια ε, κοιτάξτε κοιτάξτε, σα πω, έχω χρησιμοποιήσει κάθε ποσοτικό μέσο είχαμε στη διάθεσή μα και όταν δεν υπήρχαν ποσοτικά δεδομένα, τότε στηριχθήκαμε σε ποιοτικά δεδομένα, ανεγνωρισμένα μάλιστα από την μονάδα Impact Assessment του Κοινοβουλίου, του ίδιου. Και όπου είχαμε στηριχθεί σε ποσοτικά δεδομένα. καταρχά τα δημοσιεύσαμε και δεύτερον ε, εξηγήσαμε πώς έγινε ο υπολογισμός τους για το κόστος ε, των συναλλαγών. Δεν υπάρχει οριστικός ορισμός, σε παραδείγματι, στον οποίο να μπορούσαμε να στηριχθούμε και αυτό πάλι στηρίζεται στην... και αναγνωρίζεται από τη δική σας ε, μονάδα αξιολόγησης συνεπειών. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι αυτό που αναφέρατε ως προς την ύπαρξη διαφορετικών μοντέλων και εδώ κυρία Γκέπχαρτ μιλάμε για την ελάχιστη εναρμόνιση και αυτή θέλουμε να εφαρμόσουμε εναντί τη πλήρους εναρμόνισης. Η ελάχιστη εναρμόνιση παρουσιάζει τα εξή προβλήματα όμως, ότι δεν επιτυγχάνει τον στόχο της κατάργησης των διαφορών μεταξύ των εθνικών ε, ε, νομοθεσιών, γιατί θα παραμείνουν ενισχύει οι εθνικές νομοθεσίες, και τόσο η ελάχιστη όσο και η πλήρης εναρμόνιση παρουσιάζουν το εξή πρόβλημα ότι οι επιχειρήσει οι οποίε δεν θέλουν, δεν ενδιαφέρονται να εξαγάγουν, ότι θέλουν να δραστηριοποιούνται μόνο στο εσωτερικό, πάλι θα επιβαρυνθούν με τα ε, τέλη εκείνα τα οποία προβλέπονται ε, για να εξοικειωθούν με την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν το κόστος θα υπάρξει στην περίπτωση του δυνητικού συστήματος ε, μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέξουν το δυνητικό σύστημα, πολύ χαμηλότερο κόστος ως εκ τούτου και άρα πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο ε, υπερσυνοριακά. Και ήθελα στην κυρία Γκέπχαρτ να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι πάει κάποιος σε ένα κατάστημα να αγοράσει ένα προϊόν. Το αγοράζει με βάση το εθνικό του δίκαιο. Ή έχει το iPad στα χέρια του, κοιτάει στο διαδίκτυο, ψάχνει να βρει μια καλύτερη προσφορά από έναν ε, πολιτή που είναι εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος και άρα βλέπει ότι είναι και φθηνότερο το προϊόν. Ο κοινό καταναλωτή, και το έχουμε δει αυτό από όλε τι έρευνε που έχουμε κάνει, έχει. Γιατί έχουμε κοιτάξει ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία προχωρεί σε μια συναλλαγή. Τιμή και αξιοπιστία του ε, πολιτή γιατί δεν ενδιαφέρεται να κοιτάξει αν υπερσυνοριακά ισχύει διαφορετικό ε, νομοθετικό πλαίσιο ή όχι. Δεν γνωρίζει, διαβάζει σπάνια τις γενικές συνθήκες πολίσεων και αν τις διαβάσει πάλι δεν καταλαβαίνει και τι λένε. Άρα λοιπόν αποφασίζει με βάση τον πολιτή, την, την μάρκα δηλαδή και την τιμή. Και άρα εκεί μπορεί να υπάγεται ε, ωραιότατα ένα προϊόν στο ευρωπαϊκό ε, με βάση το Ευρωπαϊκό Καταναλωτικό Δίκαιο σε μια προσφορά τιμής πιο φθηνή, πιο οικονομική, με προστασία καταναλωτού, αντίστοιχη με αυτή του κοινοτικού κεκτημένου και μη εναρμονισμένων εθνικών δικαίων. Δηλαδή έχει ένα οικονομικό πλεονέκτημα με μεγαλύτερη προσφορά, χαμηλότερες τιμές, αφενός χωρίς να κινδυνεύει σε τίποτα ε, ε, ως προς τη νομική του, στα δικαιώματά του. Και κάτι ακόμα που είπε ο κύριος Κρότσμαν. Δεν χρειάζεται να πάει να ψηφίσει, να, να αγοράσει από το ίντερνετ ο καταναλωτή. Δεν είναι υποχρεωμένο δηλαδή να το πράξει. Γιατί μπορεί να μένει στο κατάστημα στο οποίο βρίσκεται και να πει ότι να δεν με ενδιαφέρει η τιμή τόσο πολύ ή κάτι άλλο, κάποιο άλλο μέλημα, αλλά έχω εμπιστοσύνη στον καταστηματάρχη, στον πολιτή μου και το προϊόν με ικανοποιεί και θα το αγοράσω με βάση το εθνικό δίκαιο. Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν παραβιάζει τις αρχές της Ρώμης 1. Και επίσης, για να ολοκληρώσω, τελευταίο σημείο, για να απαντήσω πολύ στο μας τον κύριο Φόξ στα αγγλικά. Πολύ... Με, ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά που είπατε για τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν για τις τροπολογίες ελάχιστης εναρμόνισης κάποιων ε, ευρωβουλευτών. Με βάση τον κώδικα δικαιοντολογίας, κάθε νομίζω θεσμικό όργανο ελέγχει εάν θα προτείνει αλλαγέ Φερρυπίν, στην μελέτη αντικτύπου. Εμείς την κάναμε. Είναι πολύ εκτεταμένοι, είμαστε περήφανοι και ήταν και πολύ καλή και ευχαριστώ πρόεδρε. right. well, we, we Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώσουμε αυτό το σημείο. Προφανώς οι συγητέ πρέπει να δουλέψουν ακόμα περισσότερο για να ετοιμάσουν ε, δύο, διαφορετικού διαφορετικούς καταλόγους Ε, δεν ήθελα να ξανακάνουμε τη συζήτηση που έχουμε ήδη κάνει, ούτως ή άλλως εκτεταμένα. Από αυτά που είπαμε όμως, ε, φαίνεται ότι η Κομισιόν αδυνατεί ακόμα να πείσει πολλούς ανθρώπους για την ορθότητα της πρότασής της και αυτό το δείξει ψηφοφορία, εν πάση Τώρα θα έχουμε δύο διαφορετικές θέσεις με τις τροπολογίες και οι δύο εισηγητές θα πρέπει να ετοιμάσουν τον κατάλογο ψηφοφορία να ψηφίσουν να τον ετοιμάσουν. Και θα πρέπει στις 17 και 18 Ιουνίου, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε τις συμβαστικέ τροπολογίες. Τώρα, αν τα καταφέρετε ή όχι, δικό σας θέμα, αλλά είναι σημαντικό να συζητήσουμε τους συμβασμούς και πώς θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Την επόμενη φορά, λοιπόν, θα πρέπει να συζητήσουμε τη στρατηγική ψηφοφορία και τις δύο εναλλακτικέ που προκύπτουν, ούτω ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν και οι βουλευτέ τι προτιμούν και θα ψηφίσουν. Και αν μετά υπερισχύσει η άποψη τη κυρία Γκέπχαρντ, μπορούμε να ζητήσουμε και άλλη μελέτη αντικτύπου. Υπάρχουν μελέτε αντικτύπου με τι οποίε διαφωνούμε. Αλλά πέρασε ο χρόνος για να ληφθεί απόφαση για μελέτη αντικτύπου. Το τι θα κάνει τώρα η, Ιρλανδική Προεδρία και η Λιθουανική Προεδρία είναι θέμα του Συμβουλίου. Αυτοί θα αποφασίσουν τι προτεραιότητα θα δώσουν. Άκουσαν τα σχόλια και του κυρίου Φόξ και τη κυρία Κέπχαρτ για αυτό το θέμα, ούτω ή άλλω η πρόσωπη τη Ιρλανδική Προεδρία. Και τώρα, αν δεν θέλουν οι εισηγητέ να επανέλθουν, λέω να κλείσουμε αυτό το σημείο. Θα ξανασυζητήσουμε αυτό το σημείο στι 17 και 18 Ιουνίου για το πώ θέλετε να προχωρήσετε με τι τροπολογίε. Ούτω ή άλλω ήταν ασύνηθη, ασυνήθιση συζήτηση που κάναμε ήδη. Ευχαριστώ τους εισηγητές και ευχαριστώ και την, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τα κατάφερε να έρθει. Ε, και τώρα η αίθουσα γεμίζει με καπνό. Για να το πω πιο, καλά, με ειδικού του καπνού, όχι με προϊόντα καπνού. Uh, now, um, um, Παρακαλώ, ησυχία. Γιατί πρέπει να περάσουμε κατευθείαν στη συζήτηση. Στο θέμα μας, το επόμενο. Έχουμε πολλές τροπολογίες για την οδηγία προϊόντων καπνού. 481 τροπολογίες ασχολείται η συγκήτρια, η κυρία Χάνσλικ, η κυρία Στάιλερ είναι εδώ, από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Κρόιτσμαν. Παρακαλώ, προσέξτε με. Εκπροσωπείται τον κύριο Σμιτ ή θα έρθει ο κύριος Σμιτ. Ο κύριος Σίνστραμ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μπίντεν δεν είναι εδώ. Ίσως ξανάρθει. Πάντως, ναι, μάλλον θα ξανάρθει. Δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ πάντως. Και ποιο εκπροσωπεί την Επιτροπή για αυτό το θέμα. Ο κύριος Ρης. Όχι, γνέφει η Επιτροπή. Ποιος είναι ο υπεύθυνο για τα θέματα καπνού από πλευράς Κομισιόν. Ο κύριο Νίσελ ή Σνίτσελ ή Σνίκελ. Μπορείτε να πείτε εσεί το όνομά καλύτερα γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Ο κύριο Σνίκελς είναι τμήματάρχη για τον έλεγχο προϊόντων καπνού και θα σχολιάσει τα, τις τροπολογίες αργότερα. Και θα ακούσει και το Συμβούλιο σίγουρα πολύ προσεκτικά. Κυρία Χάνσλικ, ποιε είναι οι απόψει για αυτέ τι 481 τροπολογίε, πέρα από το γεγονό ότι είναι υπερβολικά πολλέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Φυσικά, όπως είπε και ο Πρόεδρος μας, ο Μάλκολμ Χάρμπορτ, υπευλήθησαν για την γνωμοδότηση αυτή 481 τροπολογίες. Με χαροποιεί το γεγονός ότι αφορούν πολλούς τομείς για τους οποίους ήδη διαφαίνεται δυνατότητα συμβαστικών τροπολογιών. Βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα που είναι πιο επιμέχα και δημιουργούν περισσότερες προκλήσεις. Ας ξεκινήσω από τα πλούστερα θέματα, από τα ευκολότερα. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, οι περισσότερες τροπολογίες αφορούν τη διαγραφή των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και υπάρχει συμφωνία γιατί θεωρούμε ότι η αρμόδιότητα για την ε, μέγιστη περιεκτικότητα στο προϊόντα καπνού θα πρέπει να επαφηθεί στους ε, νομοθέτες, στους συνομοθέτε και όχι σε τη πράξη. Δεν έχουμε πρόβλημα με το άρθρο αυτό. Το άρθρο 5. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες προκειμένου να συμπεριληφθεί η υποχρέωση καταγραφή και των νοικοτινούχων προϊόντων καθώ και φυτικών προϊόντων καπνού. Επίσης, η διαγραφή της υποχρέωσης δήλωσης ε, κάποιων ε, θεμάτων σε ό,τι αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απλούστευση. Επίσης, υπάρχουν τροπολογίες σε ό,τι αφορά την εξαίρεση κάποιων προϊόντων καπνού όταν δεν αφορούν τα, το καπνό και στεφτά τσιγάρα, τσιγάρα και τα σιγαρέτα. 175, 176 και 177 είναι οι σχετικές τροπολογίες. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το ποια θα πρέπει να είναι η θέση μας απέναντι στο άρθρο αυτό. Το επόμενο άρθρο είναι το άρθρο 12. Για το άρθρο αυτό έχουν κατατεθεί πολλοί άριθμες τροπολογίες, αφορούν την περιγραφή των προϊόντων. Υπάρχουν και τροπολογίες ε, που ζητούν διαγραφή για την, το χαρακτηρισμό σιγαρετών. Συμφωνώ με το άρθρο 12, όπως το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρώ ότι στη συσκευασία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία που παραπλανούν τον καταναλωτή ή που δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι λιγότερο επιβλαβές το προϊόν. Παρ' όλα αυτά, η, το πάχος, η διάμετρος ε, του τσιγάρου δεν είναι παραπλανητική, ε, αλλά η διαφήμιση σχετική μπορεί να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Έχουμε και καταναλωτές όμως που είναι πολύ καλά κατατοπισμένοι και ενημερωμένοι, οπότε αυτοί θα πρέπει να έχουν επιλογή. Γιατί αν δεν υπάρχει τέτοια επιλογή θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα πολύ χοντρά τσιγάρα ή τα πουρα. Αλλά κανένας δεν προτείνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πληροφορίες στη συσκευασία και οι προειδοποίησεις για την υγεία έχουν κεφαλαιώδη σημασία, αλλά η διάμετρος των σιγαρέτων μπορεί να είναι διαφορετική. Στο μέτρο φυσικά που ε, θα συσκευάζονται σε χαρακτηριστικό στο, στο, στο τυποποιημένο πακέτο. Γιατί άσχετα με τη διάμετρο τα σιγαρέτα είναι εξή, θα πρέπει να τα απαγορεύσουμε όλα, είτε όχι. Αλλά η διάμετρο δεν έχει σημασία. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14, που αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα για συμβαστική τροπολογία. Όλες οι τροπολογίες αφορούν κυρίως ε, την ε, εξασφάλιση ε, καλύτερου και αποτελεσματικότερου ελέγχου των ε, ε, προϊόντων καπνού και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου τέτοιων προϊόντων. Θέλουμε να υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση, να μην είναι δυνατή η ε, να μην είναι δυνατό ο παραπλασιασμός, οπότε είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τέτοιε τροπολογίε. Τώρα, η τρίτη πλευρά που ε, ε, κρατάει τα στοιχεία σε ό,τι αφορά συγκεκριμένο παραγωγό ή εισαγωγέ, θα πρέπει αυτή η τρίτη πλευρά να είναι ανεξάρτητη, απόλυτα ανεξάρτητη από τον εμπορικό κλάδο. Και σχετικές τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Ένα άλλο όχι ιδιαίτερα επίμαχο θέμα αφορά το άρθρο 16 για την διασυνοριακή πώληση εξ αποστάσεως. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή η πλειοψηφία των τροπολογιών τάσεται υπέρ της απαγόρευσης τέτοιων πωλήσεων εξ αποστάσεως, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να εξακριβωθεί η ηλικία του αγοραστή. Επίσης ζητούμε και απαγόρευση της ε, της, παρα, της ε, προσφοράς φθηνότερων τσιγάρων ή δωρεάν τσιγάρων. 191. Επίσης ε, υπάρχει και η τροπολογία που αφορά την απαγόρευση εμφανών σημείων πωλήσεων καπνού. Νομίζω ότι η τροπολογία αυτή είναι υπερβολική. Θα προτιμούσα ε, στις ε, συσκευασίες να περιλαμβάνονται οι προειδοποιήσεις της υγείας. Θεωρώ ότι οι προειδοποιήσεις αυτές στη συσκευασία έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δεν είμαι λοιπόν υπέρ της ε, τροπολογίας αυτής που είναι πολύ πιο φιλόδοξη και υπερβολική. Επίσης, υπάρχει το θέμα των οικοτινούχων προϊόντων. Εδώ έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στις διάφορες τροπολογίες. Μερικοί ζητούν τη συμπερίληψη όλων αυτών των νοικοτινούχων προϊόντων στην οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι μερικοί ζητούν το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας να καλύπτει μόνο προϊόντα νοικοτινούχα που έχουν ε, φαρμακευτικό σκοπό. Οπότε, αν συμπεριλάβουμε στην οδηγία αυτή τα νοικοτινούχα προϊόντα, είναι σαν να τα ε, καλύπτουμε με την οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Εκεί θα πρέπει να δούμε το θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Ε, εγώ θεωρώ ότι τα πρόσωπα που θέλουν να ε, εγκαταλείψουν το κάπνισμα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή ε, και δοκιμασμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια έμπλαστρα για την απαγόρευση του καπνίσματος και άλλα νοικοτήνοχα προϊόντα και υπάρχουν σχετικέ τροπολογίε για το θέμα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και τα επιχειρήματα των καταναλωτών που λένε ότι δεν χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα για να σταματήσουν το κάπνισμα, αλλά ως καταναλωτικό προϊόν που απλώς το χρησιμοποιούν για την απόλαυση, για απόλαυση, όχι για να σταματήσουν το κάπνισμα. Ε, οι πράσινοι έχουν ε, υποβάλει τροπολογίες που ζητούν ε, ένα παράρτημα με συγκεκριμένους κανόνες για τους καταναλωτές που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Επίσης έχουμε πολλές τροπολογίες που αφορούν την μεταβατική περίοδο και ζητούν με παράταση της μεταβατικής περίοδου. Είμαι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Αυτά ήταν τα πιο εύκολα και τα λιγότερα επίμαχα σημεία, τα πιο απλά. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στα πιο περίπλοκα σημεία και τα πιο επίμαχα και να επισημάνω δύο κύριο σημεία. Το πρώτο αφορά το άρθρο 6, τα συστατικά. Ε, υπάρχει μια τροπολογία που μιλά για πλήρη απαγόρευση όλων των πρόσθετων. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες τροπολογίες που επιτρέπουν να προβλέπεται εξ, εξαίρεση για τα παραδοσιακά πρόσθετα ε, κυρίως αυτά που ε, χρησιμοποιούνται από πιο ηλικιωμένους καταναλωτές. Βέβαια, ε, υπάρχουν ακραίες όπως βλέπετε προσεγγίσεις και θα ήταν ίσως δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για το άρθρο αυτό. Αν και εγώ θα επιχειρήσω να υποβάλω συμβαστικέ τροπολογίε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρόσθετα όπως καφέινη, ταυρίνη, βιταμίνες είναι πρόσθετα που μπορούν να ενθαρρύνουν ή να παροτρύνουν τους νέου να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Οπότε τέτοιου είδου πρόσθετα ε, θα πρέπει να απαγορεύονται. Απ' την άλλη πλευρά, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει επιλογή για το τι προϊόν θα αγοράσει και θα χρησιμοποιήσει. Αν χρησιμοποιεί δηλαδή προϊόντα καπνού. Οπότε παραδοσιακά πρόσθετα που προσελκύουν κυρίως ε, πιο ηλικιωμένους καταναλωτές δεν δημιουργούν ε, πρόβλημα στην υλοποίηση των στόχων της οδηγίας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποια θα είναι η προσέγγιση που θα ώστε να περιοριστούμε σε απαραίτητη ε, τροπολογία και όχι ε, υπερβολική. Επίσης, ε, ζητείτε για το άρθρο 6, παράγραφος 10, μια εξαίρεση. Εγώ πρότεινα διαγραφή αυτής της εξαίρεσης και υπήρξαν τροπολογίες που ζήτησαν το ίδιο. Υπάρχουν όμως τροπολογίες που εμένουν στην διατήρηση αυτής της εξαίρεσης για, τις, για τον καπνό που παίρνετε από το στόμα είτε από τη μύτη. Υπάρχει ένα άλλο περιπλοκό θέμα που αφορά την ε, συσκευασία και την ετικετοθεσία. Τροπολογίες δηλαδή για τα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 13. Μερικοί ευρωβουλευτές ε, πρότειναν να μην, να, περιοριστεί, ή, ε, να μην περιοριστούν οι ελάχιστες διατάξεις των προειδοποιήσεων της υγείας. Υπάρχουν τροπολογίες που μιλάνε για ποσοστό εμφάνιση αυτών των προειδοποιήσεων. Μερικοί ζητάνε 40% της επιφάνειας, άλλοι 50%, μερικοί 50, 75%, ακόμη και 85% της επιφάνειας της συσκευασία να καλύπτεται από τις προειδοποίησεις υγείας. Επίσης υπάρχει και η πρόταση για το plain package, δηλαδή ενιαία συσκευασία. Επίσης υπάρχει περιορισμός, πρόταση για περιορισμό είτε στο άνω είτε στο κάτω μέρος του πακέτου. Άλλες τροπολογίες ζητάν διαγραφή της πρότασης για τη μορφή του πακέτου. Ενώ άλλες τροπολογίες μιλούν ε, ε, είτε για τη σακούλα που θα πρέπει να είναι, έχει οβάλ, οβάλ μορφή ή να προτείνουμε και τον τρόπο ανοίγματο τη σακούλας με το flip top. Όπως βλέπετε, οι τροπολογίες ε, βαίνουν προς πολλές και διάφορες κατευθύνσεις και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο για μένα να βρω δηλαδή μια συμβαστική λύση μεταξύ τόσο διεστάμενων ε, και διαφορετικών τροπολογιών. Γι' αυτό και περιμένω με ανυπομονησία τις θέσεις σας για το θέμα αυτό. Τέλος, ε, ε, υπάρχουν ε, πολλές και διάφορες τροπολογίες. Δεν μπορώ να σας τις παρουσιάσω όλες με λεπτομέρειες. Εγώ περιορίστηκα στην παρουσίαση των πιο σημαντικών τροπολογιών. Υπάρχει ε, διάσταση απόψεων μεταξύ των συναδέλφων. Γι' αυτό και η σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών θα είναι μεγάλη πρόκληση για την εισηγήτρια. Εγώ όμως είμαι εκφύσεως αισιόδοξη και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό θα κατορθώσω να βρω συμβαστικέ τροπολογίε για τα σημεία που σα προανέφερα. Πάντω είμαι πρόθυμη και συνεργατική, περιμένω τι προτάσει σα και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι παρά την προθυμία και το συνεργατικό πνεύμα μου, θα είναι για μερικά θέματα δύσκολη η αναζήτηση συμβαστικών τροπολογιών και για μερικά θέματα θα πρέπει ίσως να παραιτηθούμε από ορισμένε απαιτήσει μας για να κερδίσουμε κάποιες άλλες. Θα πρέπει να είμαστε ενδοτικοί και υποχωρητικοί σε διάφορα θέματα. Περιμένω λοιπόν τα, σχόλιά σας, τα σχόλιά σας, γιατί επαναλαμβάνω η γνώμη σας θα είναι πολύ σημαντική και πολύ χρήσιμη για να διαμορφώσω συμβαστικέ τροπολογίες μαζί με τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Well, thank you very much for your very clear analysis of all the amendments, which I think was extremely... Σας ευχαριστώ για την πλήρη αυτή ανάλυση. Ας ακούσουμε τους κοιόδης εισηγητές οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα θέλουν να υπερασπιστούν τις δικές τροπολογίες. Η κυρία Στάιλερ, καταρχήν, ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω και εκείνη και το γραφείο της. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην υποστηρίζετε, κυρία ε, Χάντζλικ, την, α, ε, τις τροπολογίες της ομάδας μου, αλλά ελπίζω να φτάσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες που να μπορεί τουλάχιστον να υποστηρίξει και η σοσιαλιστική ομάδα. Ας ε, ξεκινήσω με τις πιο προβληματικές. Ε, η απαγόρευση της ε, διασυνοριακής πώλησης τσιγάρων. Μ' αρέσει αυτή. Αλλά θα πρέπει να σταματήσουν και οι διαφημίσει των σημείων πώληση. Ε, το χάρη, τα έχουμε εισαγάγει στη Σκοτία πολύ εκτεταμένα και νομίζω ότι κάνει διαφορά. Είναι γνωστό ότι η διαφήμιση ε, χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η πώληση των ε, προϊόντων του καπνού. Και η διαφήμιση των σημείων πώληση είναι πάρα πολύ σημαντική. Επηρεάζει πάρα πολύ τους άμεσους, τους νέους και το 2006 46% των ε, νέων του Ηνωμένου Βασιλείου ήξεραν πολύ καλά πού πωλούνταν τα τσιγάρα. Και εκείνοι που θέλουν να καπνίσουν θυμούνται μάρκες που έχουν δει στα σημεία πώληση. Και στην Νορβηγία ε, βλέπουμε νέους πιο συχνά στα καταστήματα ε, να ψάχνουν προϊόντα καπνού από πιο ηλικιωμένους. Επομένως είναι σημαντική αυτή η απαγόρευση. Επίσης καλή απαγόρευση τη, της ε, δωρεάν διάθεσης ε, προϊόντων καπνού, τσιγάρων ή α, τσιγάρα με έκπτωση. Είναι πολύ σημαντική η ιδέα αυτή. Όμως, με ανησυχεί η τροπολογία για τα τσιγάρα μέντας και η, η ένδειξη ότι δεν, η υπονόηση ας πούμε ότι δεν είναι τόσο επιβλαβή. Έχουμε ακούσει ένα γερμανικό κέντρο να μας λέει πόσο επιζήμια είναι αυτά τα τσιγάρα μέντας γιατί καλύπτει τη μυρωδιά του τσιγάρου και διευκολύνει την απορρόφηση, αυξάνει λοιπόν τον κίνδυνο του καρκίνου γιατί εισπνέει πιο βαθιά. Τότε αυξάνει ο κίνδυνος ε, καρκίνου. Ε, επίσης, πολλοί λένε ότι αυτή ότι δεν, είναι, δεν είμαστε εμεί ε, υπεύθυνοι για την ε, υγεία του καταναλωτή. Λένε λάθο αυτό. Είναι παραπλανητική διαφήμιση, άρα δεν μπορώ να υποστήριξω αυτή την ε, τροπολογία. Σε ό,τι αφορά τη συσκευασία. Εγώ ζήτησα απλέ συσκευασίε. Καταλαβαίνω όμω ότι ορισμένε ομάδε ε, θεωρούν ότι είναι υπερβολικό αυτό. Παρότι είδαμε πόσο επιτυχή είναι αυτή η προσπάθεια σε άλλε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν για μένα οι προειδοποίησει υγεία στο πακέτο είναι κάτι που πετύχαμε στις προηγούμενες ε, διαπραγματεύσεις το 2002 ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Προειδοποίησης για την υγεία. Τώρα, η, αποδυνάμωση α, από το 75% στο 50% της επιφάνειας της συσκευασία δεν το δέχομαι. Σε ό,τι αφορά τι ε, συνολικά τι τροπολογίε, ανησυχώ γενικά ότι υπάρχει μια προσπάθεια να περιοριστούν τα δικαιώματα των κρατών μελών να πάνε πιο πέρα από την οδηγία. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την ενιαία αγορά για να κρατήσουμε πολύ χαμηλά τα πρότυπα, μόνο και μόνο προ όφελο τη καπνοβιομηχανία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία αγορά ε, ει βάρο τη υγεία ε, των πολιτών. Προς το παρόν ε, φαίνεται ότι οι θέσεις μας σε πολλά ζητήματα είναι αντιδιαμετρική. Παρόλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Χάνσλικ που έχει ανοιχτό χαρακτήρα, μπορεί να την πλησιάσει κανείς εύκολα, είναι προσίγωρη και πιστεύω ότι θα τα βρούμε σε κάποιο βαθμό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προσπαθίες σας και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Στάιλερ, ο κύριος Κρόιτς, εκ μέρους του κύριου Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να είναι κανείς σκιώδη στην, στην Ήτρε. Έμαθα από συνάδελφο των σοσιαλιστών ε, ότι να μου λέει κάποια άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά από αυτά που άκουσα από την κυρία Στάιλερ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, γιατί βλέπω ότι έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις εδώ μέσα στην Επιτροπή ας πούμε, Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Ήτρε, οι απόψεις είναι τελείως διαφορετικές. Θέλω να σας πω τι, θέλει να... τι απόψη θέλει να περάσει ο κύριος Όλη Σμιτ. Ευχαριστεί την εισηγήτρια για τις... και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστεί που και οι δικές του να λαμβάνονται υπόψη, ε, που οι εξαιρεσει ε, για το σουηδικό σνούς ε, για τα πακέτα κτλ. συμπεριλαμβάνονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους Σουηδούς. Και το ακούσαμε και αυτό και στην Επιτροπή Ήτρε. Ωραία αυτό. Υποστηρίζει τον, τους συμβιβασμούς για την ανιχνευσιμότητα και τις περισσότερες τροπολογίες γενικά μπορεί να τις υποστηρίξει. Έχει λίγες ανησυχίες, δεν τις αναφέρει όμως, άρα σας λέω μόνο τα θετικά. Θα τις δώσω ιδιωτικά στο, στην εισηγήτρια. Επίσης, για τη μέντα, τσιγάρα μέντας, αυτό μπορεί να δημιουργήσει, η εξαίρεση αυτή μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίε στους καταναλωτέ και στις επιχειρήσει για το αν επιτρέπονται τελικά τα αρώματα ή όχι. Ε, προς, θα περιμένει το συμβιβασμό. Ο στόχο τη οδηγία είναι να παρεμποδίσει τους νέου να αρχίσουν το κάπνισμα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε περισσότερα προγράμματα. Στη χώρα μου, στη Γερμανία, έχουμε πολλά και μεγάλα προγράμματα και έχουμε προχωρήσει πολύ χάρη σε αυτά τα προγράμματα. Τα νούμερα δείχνουν ότι έχουμε μειώσει το κάπνισμα των νέων. Αν το πετύχει αυτό, ε, τότε εξασφαλίζει την υγεία των μελλοντικών καταναλωτών. Γιατί νέοι είναι μελλοντικοί καταναλωτέ. Είναι σημαντικό για την παιδεία του, αλλά και το πιο σημαντικό για μένα είναι οι γονεί, δηλαδή το σπίτι του, εκεί που ζουν ε, οι νέοι, να μην καπνίσουν κι αυτοί. λεπτά τσιγάρα. Μπορεί να είναι παραπλανητικά, λέει ο Λεσμίτ. Θα προτιμούσε την πρόταση της Κομισιόν από αυτόν. Δεν είναι υπέρ τη απαγόρευση των διασυνοριακών εξαποστάσεων πωλήσεων, αλλά συμφωνεί ότι είναι δύσκολο θέμα. Ε, είναι έτοιμος όμως να συνταχθεί με την πλειοψηφία προκειμένου να βρεθεί συμβασμό. Αυτά που ήθελε να πει όλα και όλα ο Λεσμίτ και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιέλλαν που έρθει, είχε έρθει στο μεταξύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την γνωμοδότηση της κυρίας ε, Χάνσλικ ουσιαστικά έχουν κατατεθεί σχεδόν 500 τροπολογίες και σίγουρα η κατάρτιση βαστικών τροπολογιών θα απαιτήσει γιγαντιαία προσπάθεια από πλευρά της και φυσικά μεγάλη συνεργασία στην Επιτροπή. Εγώ θα αναφερθώ στα κυριότερα σημεία των τροπολογιών μας. Καταρχήν, συμφωνώ με την πρόταση επιτροπή ότι αφορά την απαγόρευση της χρήσης προσθέτων που δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο επιβλαβής ο καπνός, ότι ε, δημιουργεί ενέργεια. Επίσης, ε, για τις ετικέτες ή ε, κάποιες πληροφορίες που μπορεί να παραπλανήσουν διαφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι το μέγεθος μπορεί να επηρεάσει ε, το, την επιλογή. Αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους προϊόντα να διαφημίζονται. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δικαίωμα επιλογή του καταναλωτή, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και σωστή ενημέρωσή του. Γιατί κάθε τσιγάρο, κάθε προϊόν καπνού είναι επιβλαβέ για την υγεία, άσχετα από τη συσκευασία του ή από τη μορφή του. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να διαλέγει κατατοπισμένος και ενημερωμένος, όχι να περιορίσουμε την επιλογή του. Επίσης, για την τροπολογία σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα προϊόντα, απαραίτητα συστατικά συμφωνώ. Σε ό,τι αφορά τα σιγαρέτα μενθόλης, αυτά κυρίως ε, καπνίζονται από πιο ηλικιωμένους καπνιστές και δεν ε, νομίζω ότι εθαρρύνουν τους νέους να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Γι' αυτό τελικά αποφάσισα να υποστηρίξω την πρόταση για εξαίρεση των σιγαρέτων μενθόλης από το πεδίο εφαρμογής οδηγία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, α, τις πωλήσει μέσω διαδικτύου, νομίζω ότι αυτό μπορεί να διευκολύνει τους ανήλικους να αγοράσουν καπνό. Γι' αυτό και συμφωνώ να απαγορευτούν τέτοιες πωλήσει από το διαδίκτυο. Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ικανογραφημένες προειδοποιήσεις ή τις προειδοποιήσεις με κείμενο. Επίσης, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές αυτές οι προειδοποίησεις, αλλά δεν συμφωνώ με το plain packet, με την απόλυτη εναρμόνιση της συσκευασίας. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικό αυτό από την άποψη της ε, ελεύθερης αγοράς. Σε ό,τι αφορά τα νοικοτινούχα προϊόντα, συμφωνούμε με τις τροπολογίες της ηγήτριας για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι όλα αυτά τα νοικοτινούχα προϊόντα θα πρέπει να υπάγονται στην οδηγία 80 ε, ε, ε, για τα φαρμακευτικά προϊόντα και πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέπετε για τα προϊόντα αυτά ελάχιστο όριο ηλικία για τη δυνατότητα αγοράς. Θα ήθελα να πω ότι αναφέρθηκαν πολλές τροπολογίες για το άρθρο 13 δεν κατάφερα ακόμη, δεν πρόλαβα να τις εξετάσω όλες. Πιστεύω όμως θα πρέπει να επιτρέψουμε κάποια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τη συσκευασία διαφόρων προϊόντων καπνού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το την ποσότητα των σιγαρέτων προτιμώ τη λιγότερη δυνατή ποσότητα γιατί όσο ε, περισσότερα ίσως σιγάρι υπάρχουν στο πακέτο τόσο πιο εύκολη θα είναι η πρόσβαση για τους ε, ανήλικους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Um, να δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να μας πει την άποψη έχει για τις ε, τροπολογίες και συνεχεία θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Χάντλικ για να μας πει τι θα κάνουμε στο μέλλον. Α, κυρία Ρόιτοβα, πω, πω, πω, σας ξέχασα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν σας θωνώ, κυρία εισηγήτρια. Δεν θωνώ ότι το έργο σας είναι τόσο δύσκολο, τόσο βαρύ. Ε, έχετε τόσες πολλές τροπολογίες που είναι αντιφατικές μεταξύ τους, που σίγουρα θα μας διαρέσουν και κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, είμαι γιατρός και Επομένως θα σε εκπλήξει το γεγονός ότι έχω ξεκάθαρες απόψεις για τον κανονισμό αυτό. Για το τι θα πρέπει να ρυθμίζει και τι όχι. Και ως μέλος της Επιτροπής ΙΜΚΟ πιστεύω ότι όλες οι παραπλανητικές ε, δηλώσεις, όλες οι διαφημίσεις θα πρέπει να διαγραφούν. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Ο βασικός στόχος και συμφωνήσαμε να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα. Απλά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επομένω, το... η πορεία που έχει ακολουθεί η Κομισιόν είναι η ότι Θέλει να αποθαρρύνει τους νέους ε, να αρχίσουν το κάπνισμα. Δεν είναι εύκολο να επηρεάσουμε τους μακροχρόνια καπνιστές. Δεν είναι εύκολο έχουν την άποψή τους. Δεν μπορούμε να τους επηρεάσουμε με το μέγεθος των προειδοποιήσεων, με τη συσκευασία και με όλα αυτά τα θέματα. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να αποθαρρύνουμε τους νέους να αρχίσουν να καπνίζουν. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα τσιγάρα τα λεπτά, τα slim. Γιατί δίδεται η εντύπωση ότι α, δεν είναι και τόσο βλαβερά, γιατί είναι μικρούλια Εγώ πιστεύω ότι τα τσιγάρα δεν θα πρέπει να είναι ελκυστικά. Θα πρέπει να έχουν την ίδια όψη ό,τι και να περιέχουν. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και αποτίμηση του κινδύνου, πέρα από τις προσωπικές μας ε, απόψεις και εντυπωσει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις επιστημονικές γνώσεις στη συζήτηση. Η συζήτηση δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων στο πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Υπάρχει και το εντυπωσιακό παράδειγμα της Αυστραλίας. Η απόφασή τους όμως ήταν πιο εύκολη εκεί, στην Αυστραλία. Εδώ έχουμε 27 κράτη-μέλη που πρέπει να συμφωνήσουμε. Ενώ η Αυστραλία είναι ένα κράτος και έχει 22 εκατομμύρια κατοίκους μόνο. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά, εν υπάρχουν μελέτε και το ερώτημα είναι αν αυτέ οι μελέτε είναι αντικειμενικέ ή αν από πίσω υπάρχει κάτι. Επιδιώκουν κάποιο στόχο. Αν είναι ουδέτερε δηλαδή. Η Κομισιόν θα πρέπει να μα πει ποιε είναι οι πηγέ που χρησιμοποίησε. Γιατί πιστεύει η Κομισιόν ότι το α ή το β αυξάνει την ελκυστικότητα του τσιγάρου, ε, η τάδε ουσία είναι πιο επιζήμια από την άλλη. Πρέπει να τα ξέρουμε όλα αυτά. Πρέπει να ξέρουμε τι επιστημονικέ πηγέ που χρησιμοποίησε η Κομισιόν. Α πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα όμω. Η βιομηχανία του καπνού ε, επενδύει στην ανάπτυξη. Και πολύ σύντομα θα έχουμε τσιγάρα που θα που θα μπορούν, που θα είναι που δεν θα έχουν όλες αυτές τις επιβλαβείς ουσίες που παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης του τσιγάρου. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι παθητικοί καπνιστές δεν θα εκτίθενται σε αυτές τις επιζήμιες ουσίες πλέον. Χάρη σε αυτές τις α, ε, επαναστατικές αλλαγές της, α, ε, των επενδύσεων της καπνοβιομηχανίας και αν αποδειχθεί βέβαια ότι αυτές οι χημικές αντιδράσεις θα πάψουν να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια τη καύση, δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να, είμαστε, να υπαγρυπνούμε, να παρακολουθούμε αυτέ τι εξελίξει. γι' αυτό υπέβαλα τι τροπολογίε μου σε ό,τι αφορά την επίπτωση που υπάρχει στου παθητικού καπνιστέ. Τέτοιε πληροφορίε λοιπόν θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μα. και θα πρέπει να τι αποκαλύπτουν αν τι έχουν και οι επιχειρήσει. Και εμεί βεβαίω θα πρέπει να παρακολουθούμε τι εξελίξει. Επίση, ξέρω ότι υπάρχουν γιατροί που συστήνουν στους ασθενείς τους, σε αυτούς που καπνίζουν πολύ, να περάσουν σε ένα άλλο είδος καπνού ή προϊόντων καπνού. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Το πώς ενημερώνονται δηλαδή οι ασθενείς, ο κόσμος γενικά, για τις επιπτώσεις του καπνίσματος και του καπνού. Φυσικά πρέπει να εξαλείψουμε τις διαφημίσεις των προϊόντων καπνού Αλλά αν είμαστε πραγματικά τόσο αυστηροί, δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τις νέες εφευρέσεις και τα νέα προϊόντα να μπαίνουν στην αγορά. Πεςτε μας, Κομισιόν. Εσείς, Κομισιόν, ενημερωθήκατε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων από τη βιομηχανία. Γιατί, λοιπόν, Κομισιόν, δεν σκέφτεται τι εναλλακτικέ λύσεις. Δηλαδή, να τεθούν στην, στο εμπόριο ε, τσιγάρα που δεν θα έχουν τις ευλαβερές ε, συνέπειες των σημερινών τσιγάρων κατά τη διάρκεια της καύσης κτλ. Και, και επίσης τι άποψη έχετε για τις, παρεμβα... για τις διαφημίσεις. Ο επόμενος συνάδελφος. Ο κύριος Μπορισόφ. Είναι περίπλοκο το θέμα που αφορά τα, την δημόσια υγεία και το δικαίωμα επιλογή του καταναλωτή σε μια πλούσια αγορά, θέσει απασχόληση που υπάρχουν στην καπνοβιομηχανία κτλ. Εξού και οι πολυάριθμε τροπολογίε. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτών των διαφόρων πτυχών και να δούμε κατά πόσο οι πρώτε Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, θα, θα υλοποιήσουν το στόχο του νομοθετικού κειμένου, δηλαδή αποτρέψουν ε, του νέου ε, να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Θα επικεντρωθώ στι δικέ μου τροπολογίε. Η πρώτη αφορά τα τσιγάρα με Κύριε Μπορισόφ, ε, παρακαλώ επιβραδύνετε λίγο το ρυθμό, γιατί διαβάζετε με πραγματικά ηλικιώδη ταχύτητα. Το πρώτο μου σχόλιο αφορά τα τσιγάρα μενθόλης. Τα τσιγάρα αυτά δεν θα πρέπει να τύχουν ίση μεταχείριση με άλλα σιγαρέτα που έχουν ε, αρώματα. Γιατί η μεθόλη χρησιμοποιήθηκε ω άρωμα για το τσιγάρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το 1924 πρώτο χρησιμοποιήθηκαν, εδώ και 90 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό άρωμα καπνό. Θα πρέπει να εξαιρείται λοιπόν να μην εμπίπτει στην γενική απαγόρευση για τα αρώματα. Άλλωστε, η απαγόρευση των σιγαρέτων μενθόλη θα έχει διπλά αρνητικά αποτελέσματα για το καταναλωτή. Θα περιορίσει την επιλογή του και θα του στερήσει προϊόντα αγαπημένα. Επίση, ε, ίσω ε, έτσι δημιουργηθεί ένα παρεμπόριο σιγαρέτων Μενθόλη που θα είναι πολύ πιο επιβλαβή. Θα πρέπει λοιπόν οι καταναλωτέ που είναι συνηθισμένοι στη σιγαρέτα μεθόλη να εξακολουθούν να μπορούν να τα αγοράζουν. Σε ό,τι αφορά τα λεπτότερα τσιγάρα, τα slims, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση ε, των σιγαρέτων με διάμετρο κάτω των 7 χιλιοστών. Δεν νομίζω ότι είναι λιγότερο επιβλαβή τέτοιου είδου λεπτά τσιγάρα. Ε, διαφορώ με την εξαίρεση, με την απαγόρευση αυτή γιατί ε, και σίγουρα η διαφήμιση είναι παραπλανητική. Θα πρέπει λοιπόν να λέμε ότι όλα τα τσιγάρα είναι εξίσου επιβλαβή, κάτι που ισχύει και για τα τσιγάρα slim. Σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή πώληση προϊόντων καπνού εξ ε, πιστεύω ότι η διασυνοριακή πώληση ε, μέσω διαδικτύου ε, ε, διευρύνει την αγορά, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για την αγορά προϊόντων καπνού, γιατί δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία του αγοραστή. Θεωρώ λοιπόν ότι προς το παρόν η απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων τσιγάρα βασιλετέρων θα πρέπει να ισχύσει. Ε, είναι πολύ σημαντική η στόχη της οδηγίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσουμε δυσανάλογα μέτρα που δεν θα έφερουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά τα αντίθετα από αυτά. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις σας. Ο κύριος Νίτσελ νομίζω έχει αρκετές ερωτήσεις δεχθεί. Καλώς ήρθατε καταρχάς και παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την συγκίτρια τους και οδησηγητές και τους λοιπούς βουλευτές για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά τους. Ο κύριος Ρης δυστυχώς ε, ήταν σε μια, βρίσκεται σε μια παράλληλη συνεδρία στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος, γι' αυτό έχω εγώ την τιμή και χαρά να τον εκπροσωπώ εδώ. Θέλω να επικεντρωθώ στα θέματα της συσκευασία των ε, λεπτών τσιγάρων, ε, των ηλεκτρονικών τσιγάρων και ίσως ε, κάτι ακόμα προς το τέλος. Καταρχάς, συσκευασία και σήμανση. Είναι σαφή τα στοιχεία για εμάς, τα επιστημονικά στοιχεία. Όσο μεγαλύτερες είναι οι εικόνες, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα φέρνουν. Το 75% είναι φιλόδοξο, αλλά, φιλόδοξη αλλά ισόρροπη προσέγγιση. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου ήδη τώρα ε, σε τρεις γλώσσες δημοσιεύουν το μήνυμα ε, την προειδοποίηση υγείας σε 65% του πακέτου της συσκευασία, αυτό που ε, έχει απαιτήσει δηλαδή το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ τούτου δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από αυτό το επίπεδο το οποίο ήδη υφίσταται ή θα ήταν απίθανο να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Η, πειραματική έρευνα από τον Καναδά μας λέει ότι το 75% δίνει σαφώς ε, καλύτερα αποτελέσματα αν υπάρχουν τώρα προτάσεις ώστε να μπορούν να βάλουν το σήμα τους, ε, το εμπορικό, οι, οι επιχειρήσεις κτλ. Φυσικά και περισσεύει αρκετό χρόνο για το εμπορικό σήμα με το 5%. Επίσης, έχουν αποδείξει ε, ως προς τη συσκευασία οι επιστημονικές μελέτες ότι το ε, ο σχεδιασμός και τα διάφορα χαρακτηριστικά ενός πακέτου μιας συσκευασία μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα των καταναλωτή ότι είναι χαμηλότερου κινδύνου το περιεχόμενο σιγαρέτο και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα slim και τις συσκευασίε που βλέπετε εδώ και που συχνά περιγράφονται ως συσκευασία κραγιών ή τα ε, διαφημιστικά εκείνα κουτιά τα οποία μία ε, καπνοβιομηχανία στέλνει σε οποιονδήποτε καταναλωτή, καταναλώτρια καλύτερα, δηλώσει ότι είναι γυναίκα και άνω των 18. Ε, αρκεί μόνο το όνομα και βέβαια στη συνέχεια ρωτάνε, ζητάνε και τα ονόματα των φιλενάδων ώστε να στείλουν και σε αυτές αντίστοιχα δωρεάν κουτιά με δείγματα. Είναι προφανές ότι απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό των νεαρών γυναικών αυτή η επιθετική εκστρατεία. Βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα ότι τα slim, τα τσιγάρα αυτά, ε, απευθύνονται, προσπαθούν να προβάλλουν την ιδέα της θηλυκότητας, της κομψότητας και ως εκ τούτου δίνουν και την εντύπωση ότι είναι λιγότερο επικίνδυνα. Δεν είναι λιγότερο επικίνδυνα, ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι λιγότερο επικίνδυνα. Με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο του 2012 καταγράφεται ότι θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα τα τσιγάρα slim από τους νέους ιδίως και ιδίως συγκρινόμενη ομάδα αυτή πληθυσμού με τον μέσο όρο. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι σημειώνεται σημαντική αύξηση των πωλήσεων των τσιγάρων Slim τα τελευταία χρόνια. Σε όγκο έχουμε αύξηση 32% από το 2006 μέχρι το 2011 σε μια χώρα η οποία παρουσιάζει φθήση εν γέννη. Και είναι ως εκ τούτου σημαντικό να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο SLIM. Ω προ την νομοθεσία τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ε, απαγόρευση των προϊόντων με ισχυρό, ισχυρή γεύση. Παραδείγματι, η πολύ έντονη γεύση μεντόλης ή ε, βανίλιας, γιατί το ξέρουμε και το επιβεβαιώνουν και οι μελέτε, οι έρευνε, ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικά τα προϊόντα αυτά για τους νέους και καθιστούν ακόμη και πιο εύκολο το να ξεκινήσει κανεί να καπνίζει. Είναι αυξανόμενη και ενισχυόμενη η τάση της βελτίωσης ε, ε, γεύσεων όπως της βανίλια της, του, σοκολάτας ή τη φράουλα, και βλέπουμε την εισαγωγή μέσα στο φίλτρο ε, κα, με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού που κατέχει στην αγορά το τσιγάρο μεντόλι σε ορισμένα κράτη-μέλη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η διαθεσιμότητα προϊόντων μενθόλης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανολόγηση πειραματισμού με τα τσιγάρα αυτά των νέων και ως εκ τούτου την έξι στο κάπνισμα. Αποτελεί δηλαδή μια πολύ πιθανή αρχή καπνίσματος για τους νέου Πολύ περισσότερο από ότι σε άλλε ομάδες ηλικίας. Μπορεί να διαστρεβλωθεί η εικόνα του καπνίσματος λόγω αυτής τη ιδιαίτερη γεύση. Και επίσης και πολύ σημαντικό, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω να μην προσπαθήσετε να αποκλείσετε κάποιες γεύσει που μπορεί να θεωρούνται παραδοσιακέ ή να είναι και παραδοσιακέ. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να κάνουν ακριβώ το ίδιο πράγμα με την ίδια πρόταση ως προς τις χαρακτηριστικές γεύσεις που έχουμε κάνει και εμείς από πλευράς της Επιτροπής και ε, πήγαν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με προσφυγή, την οποία έχασαν, διότι κανένα επιχείρημα του διεθνούς δικαίου δεν επιτρέπει να ε, έχει προτιμησιακή αντιμετώπιση η μία γεύση και όχι η άλλη. Πρέπει να έχουμε την αντιμετώπιση για κάθε είδους διαφορετική γεύση. Τέταρτη παρατήρηση, ηλεκτρονικό σιγαρέτο και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σημαντική διευκρίνηση. Γιατί φαίνεται ότι επικρατεί η παρεξήγηση ω προ το τι πραγματικά θέλουμε και τι εννοεί η πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα στην αγορά. Θέλουμε να, βοηθεί, να βοηθείτε ο καταναλωτή να σταματήσει χάρη στα προϊόντα αυτά το κάπνισμα. Δεν θέλουμε να τα απαγορεύσουμε. Αλλά θέλουμε και να είναι ασφαλή Θέλουμε να είναι αποτελεσματικά και να είναι υψηλή ποιότητα. Αυτό επιδιώκουμε. Όταν λοιπόν κοιτάμε ποιο είναι το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα πρέπει να απαντήσουμε και απαντήσαμε εμείς στα εξής σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή τα σιγαρέτα. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι αποτελεσματικά για να μπορέσει κανείς να αποδεσμευθεί από, το, από τον εθισμό στο κάπνισμα. Και τρίτον, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μετατραπούν σε πύλη εισόδου στο κάπνισμα, στον εθισμό δηλαδή, για τα νέα παιδιά. Και θα σας υπενθυμίσω μία πρόταση που είδατε πρόσφατα από τη γερμανική κυβέρνηση που έλεγε ότι 64% των παιδιών από 12 έως 14 ετών δεν είχαν καπνίσει ποτέ, αλλά είχαν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κάτι δηλαδή το οποίο στο παρελθόν μπορεί να είχε βάση ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είχε, ε, ότι χρησιμοποιούνταν μόνο για να σταματήσει κανείς να αποδεσμευθεί να πεμπλακεί από το τσιγάρο, τώρα βλέπουμε ότι δεν ισχύει πια. Και ο φόβος ότι καθιστά ένα προϊόν ελκυστικό προς τον νέο επιβεβαιώνεται. Και άρα θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ε, θα πρέπει να ε, οριστεί λοιπόν ένα καλό ρυθμιστικό πλαίσιο και καλές απαντήσεις βρίσκουμε από τη φαρμακευτική νομοθεσία για το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο. Γι' αυτό και προτείνουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο κάθε τύπου ε, με ένα επίπεδο νοικοτήνη ενώτερο από χ επίπεδο να υπαχθεί στο φαρμακευτικό νομοθετικό πλαίσιο όπου ορίζονται επίπεδα νοικοτήνης για κάθε άλλο ε, τύπο υποκατάστατου νοικοτήνης. Και έτσι αποφεύγουμε και την διακριτική μεταχείριση των λοιπόν υποκαταστάτων ε, που χρειάζεται να περάσουν από τη διαδικασία τη αδειοδότηση για τα φαρμακευτικά προϊόντα και του τσιγάρου, του ηλεκτρονικού, το οποίο με αυτή την πρόταση θα υπάγεται και αυτό στην διαδικασία τη πιστοποίηση. Ε, κάποια σύντομα σχόλια για την απαγόρευση των διαφημιστικών συσκευασιών, τα όρια ηλικία, ε, όλα αυτά μα φαίνονται πολύ καλά, μέτρα καλά, για να αποθαρρυνθεί ο νέο, να μην μπορεί να ξεκινήσει εύκολα το κάπνισμα. Πιστεύουμε όμω και βλέπουμε, για λόγου και επικουρικότητα ότι θα πρέπει να είναι σε εθνικό επίπεδο η ρύθμιση μάλλον. Ε, επίσης για τα νέα προϊόντα καπνού, τα καινοτόμα, ξέρουμε ότι βρίσκονται υπό ανάπτυξη τέτοιου είδου προϊόντα. Η ΔΕΚΑ Νοφεμηχανία μας διαβεβαιώνει ότι έχουν μειωμένη διακινδύνευση τα προϊόντα αυτά. Ε, ωστόσο, ξέρουμε και έχουμε κάνει σχετικέ ε, συνεδριάσει των οποίων τα πρακτικά βρίσκονται στου ιστοτόπου μα. Εμεί λέμε ότι ε, μπορούν προϊόντα με χαμηλότερη διακινδύνευση να μπαίνουν στην αγορά, αλλά υπενθυμίζουμε στο Κοινοβούλιο ότι έχει λάβει το 2001 την απόφαση που λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς οποιαδήποτε συγκριτική διαφήμιση η οποία μπορεί να προβάλλει ένα προϊόν ως λιγότερο επικίνδυνο από κάποιο άλλο γιατί μπορεί να παραπλανεί να παραπλανά τον καταναλωτή και μπορεί να αποτελέσει επίσης και το σημείο εισόδου για το κάπνισμα ορισμένων νέων. Για τα προϊόντα, τα προϊόντα αυτά δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολοκληρώνοντας. Ήταν πολύ εντυπωσιακή συνεργασία στο θέμα αυτό. Με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε μαζί σας για το μέλλον. Ή αδίποτε ερώτηση έχετε, πολύ ευχαριστώ να σας ε, συνδράμουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ από πλευρά μου, λέει ο κύριο Χάρμπορ, απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο πλέον, τον εξαντλήσαμε. Σα άφησα να ολοκληρώσετε γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα να ευχαριστώ και του ε, διερμηνεί που έμειναν περισσότερο. Ε, κυρία Χάντσλικ, ήταν πολύ πλήρη η συνεδρίαση και η παρουσίαση. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε τώρα. Συμβαστικές τροπολογίες θα κατατεθούν. 18 Ιουνίου προβλέπεται η προσεχή συνεδρίαση και εκεί θα υιοθετηθεί η πρόταση θα εγκριθεί μάλλον η πρόταση. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη διαδικασία της έγκρισης. Σημειώσατε ασφαλώ με μεγάλη επιμέλεια ότι είχε να πει η Επιτροπή. Ευχαριστώ τους πάντες για την ε, παρουσία τους και συμβολή του εδώ. Κλείνουμε και συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα με την συζήτηση της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλία για την παραπλανητική διαφήμιση.